Συνάδελφοι, δεν έχω ξεκινήσει τη συνεδρίαση. Θα κηρύξω την έναρξη και θα σας δώσω τον λόγο. Έναρξη της συνεδρίασης. Θα περάσουμε στο σημείο 7. Ακρόαση για την μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για, τους, για τα διεθνή κριτήρια αναφοράς την παρατηρήσή σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκ μέρους της Άλντε θα ήθελα να προσθεθεί στην ημερήσια διάταξη το αίτημα για μία ε, προσωρινή επιτροπή για την διερεύνηση της ε, φοροδιαφυγής και φοροαπάτης ε, Ιδίω στα πλαίσια τη Επιτροπή, υπό την ηγέτη τη Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ε, γιατί το θέτω εδώ, Γιατί οι πολίτε ε, ασχολούνται πολύ με το θέμα αυτό και πληρώνουν φόρου και του απασχολεί. Ε, όχι μόνο για το Λουξεμβούργο και το Luxembourg αλλά θα έπρεπε να οργανώσουμε δημόσιε ακροάσει για τέτοιου είδου έρευνε και να τα συζητήσουμε και με τον ΩΣΑ σε πιο τεχνικό επίπεδο. Οπότε, Πρόεδρε, προτείνω στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, εκ μέρου τη ομάδα των Φιλελευθέρων, να αναλάβουμε την ε, πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την πρωτοβουλία και επειδή την προηγούμενη θητεία είχαμε ασχοληθεί με τα θέματα τη φοροδιαφυγή και φοροαπάτη στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμών. Πιστεύω ότι να παραμείνουμε στην εμπροστοφυλακή συζήτηση των θεμάτων αυτών. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για την πρότασή σας. στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών θα το συζητήσουμε. Ε, εν τω μεταξύ, όπως ξέρετε, υπάρχει συζήτηση. Προβλέπετε το θέμα στην Ολομέλεια, οπότε θα τα δούμε και εκεί. Στο ανώτατο σώμα του Κοινοβουλίου. Και άλλωστε υπάρχει και μόνιμη ομάδα εργασία για τα φορολογικά, όπω ξέρετε. Περνάμε στην ακρόασή μα. Ακρόαση για το πολύ σημαντικό θέμα τη ε, αναθεώρηση ή μεταρρύθμιση για την νομοθεσία των ε, διεθνών κριτηρίων αναφορά. Καλωσορίζω του προσκεκλημένου μα. Έχουμε τέσσερι ομιλητές στις Βρυξέλλες και έναν πέμπτο με τον οποίο θα συνεννοηθούμε με τηλεδιάσκεψη από τη Μαδρίτη. Καλώς ήρθατε όλοι σας. Και ζητούμε τη δική σας συμβολή στο έργο μας για τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας ε, των διεθνών κριτηρίων αναφοράς. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε ως νέα επιτροπή την όλη διαδικασία εξ αρχής με νέο εισηγητή, νέους και όδους εισηγητές, οι οποίοι φυσικά θα λάβουν το λόγο στη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα όμως ας δώσουμε το λόγο στους ομιλητές μας και ας τους ζητήσουμε να σεβαστούν το χρόνο του πενταλέπτου για τις εναρκτήρες παρατηρήσεις τους και μετά θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής. Δίνω ευθύς αμέσως το λόγο πριν τους ομιλητές στην εισηγήτρια, την Κόρα Φαν Νίβενχόιζεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, τους σκιώδεις εισηγητές για τη συνεισφορά τους προκειμένου να διοργανωθεί αυτή η ακρόαση και σε όλους τους συμμετέχοντες. Το θέμα των ε, κριτηρίων αναφορά είναι τεράστια σημασία για του Ευρωπαίου καταναλωτέ και τι επιχειρήσει. Αλλά για να υπάρχει και εμπιστοσύνη και σταθερότητα στι χρηματοοικονομικέ αγορέ. Μετά τα σκάνδαλα και ε, του χειρισμού και τι παραποιήσει του συγκριτικού επιτοκίου Euribor, ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε κριτήρια αναφορά σε κρίσιμε περιοχέ τη οικονομία και των αγορών. Πρέπει να είναι εύρωστα τα κριτήρια αυτά και αξιόπιστα. Πρέπει λοιπόν αυτό να γίνει με κάποιο τρόπο που να είναι αναλογικός, λειτουργικός και να, υπάρχει, να υπάρχουν ίσοι κανόνες ανταγωνισμού για, όλου του για όλους τους διεθνείς χρήστες των ε, κριτηρίων αναφοράς. Η σωστή προσέγγιση θα είναι δύσκολο να εξευρεθεί. Γι' αυτό θέλουμε με τους υπεύθυνους των προτύπων, τους εκπροσώπους των benchmark και τους ε, όσου τα διαχειρίζονται να έχουμε μια επικοδομητική και διαφωτιστική ακρόαση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ας ξεκινήσουμε με τις ομιλίες αυτές καθεαυτές. Πρώτος ομιλητής, ο κύριος David Wright, Γενικός Γραμματέας του ΙΟΣΚΟ, της Διεθνού, του Διεθνούς Οργανισμού για τις Επιτροπές Αξιογράφων στην Ισπανία. Κύριε Wright, έχετε το λόγο. Mr. Wright. Κύριε Ράιτ, μας ακούτε? Μας ακούτε? Ναι. Μπορείτε να ξεκινήσετε. not verbal communication, but... Ναι, ναι. Δεν είναι λεκτική επικοινωνία μας, μας βλέπετε μόνο, αλλά ναι. Please, who can communicate with our speaker? Μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με τον ε, ομιλητή μας, να πάρει τηλέφωνο ίσως. Yes, we hear you. You can... You... Ναι, εμείς σας ακούμε. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Ναι, ναι. Μας ακούτε, ναι. Hear you. I am hearing you. Ναι. Σας ακούμε. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ράιτ. Επόμενος ο μιλητής ο κύριος Ρομπέρτος Κιάβη, υποδιευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Μάρκετ, που θα μας μιλήσει για τις συναλλαγές της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κυρίες και κύριοι της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή τη δημόσια ακρόαση στο Ευρωκοινοβούλιο. Τα κριτήρια αναφοράς μέσα στα χρόνια έχουν γίνει ένα ζωτικό τμήμα της υποδομής της οικονομίας μας. Πρόκειται για δείκτες που καθορίζουν τις πληρωμές των χρηματοοικονομικών συμβάσεων, βάσει των οποίων κανένα μέρος της σύμβασης δεν μπορεί να ορίσει το πώς ε, προσδιορίζονται οι δείκτες αυτοί. Η αξία και η αξιοπιστία τους προκύπτει από την αμεροληψία, την ε, αντιπροσωπευτικότητα και τη δικαιοσύνη που τους διέπει. Η εμπιστοσύνη στην αμεροληψία ενός δείκτη πρέπει να παραμείνει. Ιδάλλως, εφόσον διαργεί, ε, η σχέση συμβασιακή μεταξύ δύο μερών θα πληγεί εξίσου. Τα ε, επιτόκια αναφορά όπω το αιώνια και το Euribor στην Ευρωζώνη έχουν γίνει ένα σημαντικό στοιχείο του διεθνού χρηματοοικονομικού συστήματο και ένα καθοριστικό εργαλείο για, την, ε, για τον καθορισμό τη νομισματική πολιτική. Η σκοπιμότητά του έχει τεκμηριωθεί από το Συμβούλιο τη ε, Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα τον Ιούλιο του 2014 στην έκθεση για, τους μεγαλύτερους, για τα σημαντικότερα επιτόκια αναφορά. Βέβαια, πολλές φορές ε, την χάνουν ε, παραποιήσεων, ε, χρησιμοποιούνται για να παραποιηθούν και να τους χειριστούν ε, προκειμένου να ε, πληγεί η εμπιστοσύνη που υπάρχει σε αυτούς. Η αποφασιστική δράση των δημόσιων αρχών θα πρέπει να είναι να τιμωρήσει την παραποίηση αυτή με μια αξιόπιστη διαδικασία που να βελτιώσει τη διακυβέρνησή τους. Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας συνεργάζονται για να επιτύχουν χειροπιαστή πρόοδο. Η σημασία της δέσμευσης του ιδιωτικού τομέα στην κοινή αυτή προσπάθεια είναι καθοριστική, διότι ο δημόσιος τομέας μπορεί να προβλέψει ένα πλαίσιο κανόνων και να στηρίξει τη διαδικασία μεταρρύθμισης. Όμως τα κριτήρια αναφοράς για τους ιδιώτες είναι κάτι που πρέπει να αποφασίζουν και να το διαχειρίζονται οι συμμετέχοντες στην αγορά. Το να ολοκληρωθεί αυτή η μεταρρύθμιση είναι κάτι βέβαια που αποτελεί ε, και επίγουσα νομοθετική πρωτοβουλία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καλωσορίζει την πρόταση κανονισμού για τους χρηματοοικονομικούς ε, δείκτες αναφοράς, όπως προκύπτει από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Σεπτέμβριο του 2013. Και ευχαριστεί το Ευρωκοινοβούλιο για το έργο εξέτασης και έγκρισης του πρότασης αυτού του κανονισμού. Ο κανονισμός ε, ορίζει την διαδικασία για την δημιουργία κριτηρίων αναφοράς προκειμένου να προστατευθεί από παραποίησεις και να προστατευτούν οι επενδυτές και οι καταναλωτές ώστε να συμπληρωθεί το νομοθετικό κενό στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον τομέα και να υπάρχουν συγκεκριμένα επιτόκια αναφοράς για την Ευρωζώνη. Η γοργή έγκριση της πρότασης αυτής από τους νομοθέτες είναι σημαντική. Ε, να θυμίσω μερικά στοιχεία από τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την πρόταση της Ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Καλωσορίζει το γεγονός η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι η πρόταση κανονισμού ορίζει ένα κοινό σύνολο εφαρμόσιμων κανόνων για, όλους, για όλη τη διαδικασία καθορισμού ε, κριτηρίων αναφοράς και για όλο το φάσμα των κριτηρίων αυτών. Εντοπίζει ποια από τα κριτήρια αυτά αναφοράς έχουν ε, συστημική σημασία, τα, ονομαζόμενα κρίσιμα κριτήρια και εφαρμόζει για αυτά ένα αυστηρότερο καθεστώς. Προβλέπεται η δυνατότητα για τη συνεργασία μεταξύ εποπτών και υπάρχει και η δυνατότητα των ε, ε, φορέων ή προσώπων που βρίσκονται υπό υποπτία να προσφέρουν πληροφορίες για τους κρίσιμους δείκτες. Έχει τονίσει επανειλημμένος η ΕΚΤ ότι η συστημική σημασία του Γιούριμπουρ για τις ε, χρηματαγορές της Ένωσης θα παίξει σημαντικό ρόλο και για τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής. Οπότε και οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές πρέπει να συμμετέχουν στην παρακολούθηση της διαδικασίας διαδικασίας ε, θέσπισης επιτοκίων. Αρχές όπω η ΕΣΜΑ και η EBA πρέπει να αναλάβουν το ρόλο αυτό ταυτόχρονα. Η ΕΚΤ ασχολείται με την λειτουργικότητα ε, του σώματος αρμόδιων αρχών για την περίπτωση των κρίσιμων δικτών εφόσον αυτό το σώμα δημιουργηθεί. Για τα επιτόκια αναφοράς, ένα φάσμα χωρών ε, θα πρέπει να συμμετέχει, όπως συμβαίνει για το Euribor. Δηλαδή ένας μεγάλος αριθμός αρμόδιων αρχών θα πρέπει να συντονίσουν τις δράσεις τους. Επιπλέον η ΕΚΤ ε, στέκεται στο γεγονός ότι το σχέδιο κανονισμού ασχολείται με τα ποσοτικά κριτήρια και αυτό ε, καθορίζει ποιοι δείκτες είναι κρίσιμοι. Όμως τα ποσοτικά κριτήρια δυσχεραίνουν την αξιολόγηση και μπορεί να μην είναι επαρκή για τα εθνικά κριτήρια που και αυτά μπορεί να, ε, θα, θα έπρεπε να ταξινομηθούν ως κρίσιμα και μπορεί να είναι κρίσιμα σε εσωτερικό επίπεδο. Επίσης, τα αριθμητικά όρια για να ζητήσουν οι επόπτες την υποχρεωτική συμβολή στα κριτήρια αναφοράς μπορεί να μην προστατεύουν τα κριτήρια αναφοράς από παρατεταμένη αλλά και βαθμιαία μείωση του αριθμού των συμβαλλόντων. Έτσι, ο ορισμός των κρίσιμων κριτηρίων αναφοράς και η υποχρεωτική συμβολή φαίνεται ότι θα πρέπει να βασίζονται και στο στοιχείο της ποιότητας. Ποιότητα που θα επιτρέπει να ληφθούν υπόψη και ε, προβληματισμοί οικονομικού και χρηματοοικονομικού περιεχομένου. Επίση, να επιστήσω την προσοχή σα στην πρόταση να δημιουργηθεί ένα καθεστώ αντιστοιχία για δείκτε τρίτων χωρών. Κάτι που θα θέλει να διασφαλίσει στου πολίτε τη Ένωση την ποιότητα των κριτηρίων αναφορά που χρησιμοποιούν και, ένα, και ισοτιμία μεταξύ όλων όσοι ασχολούνται με την ε, διαχείριση των κρίσιμων κριτηρίων αναφορά. Είναι σημαντικό αυτέ οι απαιτήσει να μην παρεμποδίσουν χωρί λόγο τη χρήση των δικτών τρίτων χωρών, επειδή είναι πολλά τα επενδυτικά προϊόντα που ε, κινούνται στην Ένωση, αλλά δεν υπόκεινται σε ευρωπαϊκά κριτήρια. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει αντίστοιχου όρου και για αυτά τα κριτήρια αναφορά και να δει τι θα γίνει με τι εκκρεμούσε συμβάσει και την, ε, τον εντοπισμό τέτοιων κριτηρίων αναφορά. Επίση, μια μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή του ε, συστήματο αντιστοιχία πρέπει να προβλεφθεί. Σε αυτήν την μεταβατική περίοδο οι υπεύθυνοι των τρίτων χωρών θα πρέπει να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους με τις διεθνείς αρχές για την θέσπιση κριτηρίων αναφοράς που εξέδωσε ο Ιώσκο τον Ιούλιο του 2013 και που είναι και η βάση για την ε, πρόταση ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το να χρησιμοποιείται ένα τέτοιο διεθνώ αναγνωρισμένο πρότυπο θεμέλιο για την αναγνώριση και το καθεστώ αντιστοιχία των δικτών των τρίτων χωρών νομίζουμε ότι είναι ιδιαίτερα εύστοχο. Να ολοκληρώσω τονίζοντα και πάλι τη σημασία του να δημιουργηθεί γρήγορα ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για τα κριτήρια αναφορά. Ο κίνδυνο για τους κρίσιμους δείκτες να καταρρεύσουν επειδή διαβρώνεται η εμπιστοσύνη των ε, συναλλασσομένων στην αγορά και όσων συμβάλλουν στην δημιουργία τους είναι ένας κίνδυνος που κανείς δεν θέλει να αναλάβει διότι θα υπάρχει τεράστιος αντίκτυπος για τους τελικούς χρήστες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Όταν δημιουργηθεί ένα τέτοιο νέο πλαίσιο θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα είναι και εύρωστο και αξιόπιστο διότι μόνο ενδυναμώνοντας την ποιότητα των υπαρχόντων και μελλοντικών κριτηρίων αναφοράς μόνο τότε θα μπορέσουμε να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη δικαιοσύνη που τους αρμόζει. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος Χάρτμον Γκράφ, εκτελεστικός διευθυντής της STOX, του Παγκόσμιου Παρόχου Δικτών. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Οίκων, ε, ε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, πρόσκλησή σας. Μεγάλο, μεγάλη τιμή εδώ πέρα να υποστηρίξω τη συζήτηση σας. Θα ήθελα να απευθυνθώ στο ερώτημα γιατί είναι τόσο σημαντικοί οι δείκτες. Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια φάση που απειλείται από την ε, Ιαπωνική ασθένεια. Δηλαδή δεν έχει ανάπτυξη, έχει πολύ χαμηλή ανάπτυξη και γυράσκει ο πληθυσμό και το indexing, η χρήση δικτών δεν πρόκειται να λύσει αυτά τα προβλήματα, αλλά ίσως να συμβάλλει σε κάποιες από τις λύσεις ε, οι επενδύσεις βάσει δικτών είναι πολύ καλύτερο τρόπος εξοικονόμησης για την ε, ε, και το 60-90% των ε, μάνατζερ δεν φτάνουν τους στόχους τους. Χρειάζονται, λοιπόν τα περιουσιακά στοιχεία που δαπανώνται, που επενδύονται σε τέτοια ταμεία να αυξάνονται. Επίσης οι δείκτες αυξάνουν και βοηθούν στην σωστή ανάπτυξη κεφαλαίου και δίνουν διαφάνεια για το τι γίνεται στην αγορά. Άρα οι δείκτες είναι σημαντικής αξίας για την οικονομία και για την επενδυτική οικονομία ιδιαίτερως. Και αυτό γίνεται με μια σημαντική προσπάθεια. Για να σας δώσω κάποια στοιχεία, έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια δείκτες στον κόσμο. Έχουμε μετοχές οι οποίες καθημερινά φτάνουν σε 120 εκατομμύρια τιμές και 30 εκατομμύρια διαφορετικές τιμές δικτών σε καθημερινή βάση υπολογίζουμε. Βρίσκομαι λοιπόν εδώ μπροστά σας ως πάροχος τέτοιων δικτών και Πιστεύω και εγώ ότι η ρύθμιση των δικτών είναι κάτι το απαραίτητο και το ωφέλιμο, γιατί η κατάχρηση τέτοιων δικτών ε, βασίζεται στη σύγκρουση συμφερόντων, γιατί αυτοί που συμμετέχουν στην αγορά και αποφελούνται οικονομικά από τους δείκτες, εμπορευόμενοι τέτοια προϊόντα που βασίζονται σε δείκτες και παροχή τιμών ε, για αυτά τα benchmark, για αυτές τις τιμές αναφοράς. Αυτή η σύγκρουση συμφερόντων λοιπόν θα πρέπει να λυθεί από την ε, νομοθεσία. Υπάρχει και μια δεύτερη σύγκρουση συμφερόντων όταν ε, ο πάροχος περιουσιακών στοιχείων ε, σχετίζει και συσχετίζει τους δείκτες με τα προϊόντα του, όπως σε κάθε περίπτωση που ελέγχονται ουσιαστικά οι τιμές και θα πρέπει να προσέξουμε από το θέμα της αυτορύθμισης βάσης δικτών. Και πιστεύουμε λοιπόν ότι χρειάζεται η νομοθεσία αυτή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά για τις περιπτώσεις κατάχρησης δικτών. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω το εξής. Χρειάζεται μια αναλογική προσέγγιση για να μην ε, υπάρξει αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, για να υπάρχουν ε, δύο μέτρα και πιο αυστηρές ε, προδιαγραφές σε ένα μόνο τμήμα του κόσμου και να υπάρχει και ένα μοντέλο επιχειρήσεων το οποίο να υποφελήσει τελικά. Δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου οι δείκτες θα υπολογίζονται από τους παρόχους προϊόντων μόνο γιατί στην περίπτωση αυτή μπορούν να επιδοτούσουν την παραγωγή δείκτων και επίσης ο αριθμός των επιλογών μειώνεται γιατί θα φεύγουν διάφοροι παροχοί από την αγορά. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε τις εξή ε, προτάσεις για μια τέτοια κανονισμό για τα κατηρία που αναφορά σύμφωνα με την αναλογικότητα. Οι απαιτήσει ε, για δείκτες βάσει ρυθμισμένων δεδομένων και ανταλλαγών δεδομένων βάσει συναλλαγών που γίνονται και οι απαιτήσει για τους δείκτες αυτοί θα πρέπει να είναι πιο χαμήλερες από τη, για τους δείκτες που έχουν να κάνουν με τις συνεισφορές στις τιμές. Δύο συγκεκριμένα παραδείγματα όπου θα θέλαμε να υπάρχει διαφοροποιημένη προσέγγιση. Καταρχάς, να μην υπάρχει καταγραφή αρχείων σε ό,τι αφορά τέτοια ρυθμιζόμενα τα δεδομένα, γιατί ήδη ρυθμίζονται τα δεδομένα αυτά, ήδη υπόκεινται στη MIFID και επίσης πιστεύουμε ότι οι δείκτες αυτής που βασίζονται σε αριθμισμένα δεδομένα δεν θα προαποτελούν μέρος των critical benchmarks, των κρίσιμων κριτηρίων αναφοράς. Η παροχή δικτών είναι παγκόσμια επιχείρηση και υπάρχει και παγκόσμιο συνταγωνισμό σε παγκόσμια κλίμακα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει και μια παγκόσμια ρύθμιση. Έχουμε Κάποιες αρχές για, τους, για τα οικονομικά κριτήρια αναφοράς ε, δημοσιεύτηκαν πέρσι και αποτελούν μια καλή βάση για μια παγκόσμια πρωτοβουλία ρυθμίσης. Αυτές οι αρχές έχουν ήδη εγκριθεί και υιοθετηθεί από τους πιο πολλούς πάροχους δεκτών και τα θέματα ισοτιμίας θα δουλέψουν μόνο αν υπάρχει ε, αναλογικότητα, αν υπάρχει ισοτιμία. Και ε, αυτό δεν γίνεται όσο η ΕΠΑ ΕΕ δεν έχει αναγνωρίσει, έχουν αναγνωρίσει τέτοιες, ε, τέτοια σωτημία. Θα πρέπει λοιπόν η ΕΕ να αναγνωρίσουν τους άλλους δείκτες και σε περίπτωση που οι αρχές των άλλων χωρών τηρούν τις απαραίτητες ε, αρχές ΑΙΟΣΚΟ. E θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η νέα ανεξάρτητη οικονομία δείκτων έχει λειτουργήσει καλά. Δεν έχουν παρουσιαστεί σκάνδαρα τις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχει προϊόντων είναι αυτή που ευθύνονται για τα σφάλματα και υπάρχει μια τελευταία ψυχή που θα ήθελα να υπογραμμίσω πριν κλείσω. Μια συζήτηση για το πώς θα βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση και τις δομές παροχής δικτών. Μια συζήτηση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ επίκαιρη για τη βελτίωση, όπως για παράδειγμα για τη βελτίωση των δημοσίων συγγενειών. Είναι πολύ σημαντική συζήτηση, αλλά φυσικά δεν θα πρέπει να γίνει συζήτηση για να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στι δημόσιε μεταφορέ. Το ίδιο ισχύει και για την ε, οικονομία των δικτών. Είναι ανεξάρτητη και ανταγωνιστική η βιομηχανία, η οικονομία. Δεν θα πρέπει να περιορίζει η ρύθμιση την λειτουργία της αγοράς ε, περιορίζοντας υπερβολικά την πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μία αναλογική, ίσως σταθισμένη προσέγγιση. Αυτές οι προτάσεις θα εξασφαλίσουν λοιπόν αυτή την ισορροπή προσέγγιση για μία ε, αγορά η οποία θα επιτρέπει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και προσβλέπω σε μία ανοιχτή και καρποφορά συζήτηση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ντεγκράφ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Ρούντολφ Ζίμπελ, που είναι πρόεδρος της ομάδας εργασίας της ΕΦΑΜΑ για τα benchmarks, τα κριτήρια αναφοράς ε, και είναι και διαχειριστικός διευθυντής του, της Γερμανικής Ένωσης Επενδυτικών Κεφαλαίων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμο κυρίες και κύριοι, ΕΦΑΜΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Περιοσιακών Στοιχείων, είναι μια αντιπροσωπευτική οργάνωση ε, που εκπροσωπεί 27 ε, ενώσεις και περίπου 17 τρισεκατομμύρια στοιχεία του ενεργητικού από τον Ιανουάριο. Θα ήθελα να πω αυτής εξ αρχής ότι ο κλάδος μου υποστηρίζει πλήρως τους στόχους του κανονισμού, γιατί θα βοηθήσει τους επενδυτές να υλοποιήσουν τους στόχους τους, κυρίως εξασφαλίζοντας εμπιστοσύνη στον κλάδο και αποκαθιστώντας τη χαμένη εμπιστοσύνη. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας διευκρινίσω το ρόλο των διαχειριστών στοιχείων του ενεργητικού διαχειρίζονται οι διαχειριστές αυτοί ως ΕΚΑ και εναλλακτικές επενδύσεις προ όφελο των πελατών που, είναι, που μπορεί να είναι είτε απλοί επενδυτές όπως εσείς εγώ είτε θεσμικοί επενδυτέ, όπως ασφαλιστικέ εταιρείε, ή ταξιδωτικά ταμεία. Ή κανονικές ε, ε, εταιρείε που χρηματοδοτούν την οικονομία. Οπότε οι, οι οικονομίες και οι συντάξεις εκατομμυρίων πολιτών εξαρτώνται από την διαχείριση των κονδυλίων των ταμείων αυτών από την ΕΦΑΜΑ. Η διαχείριση περιοχών στοιχείων από διαχειριστές δεν προϋποθέτει παραγωγή ή συμβολή σε στοιχεία που αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό των κριτηρίων αφοράς. Οι δείκτες χρησιμοποιούν το στόχο προς αναπαραγωγή ιδιαίτερα για εισηγμένα στο χρηματιστήριο κεφάλαια ή κεφάλαια που, που παρακολουθούν δίκτυ ή για την αξιολόγηση της απόδοσης ενός προϊόντος ή της απόδοσης του διαχειριστή. Επίσης δεν έχουμε πρόσβαση σε διαδικασίες θέσπισης δικτών, ούτε μπορούμε να ελέγξουμε ή να ε, χειραγωγήσουμε την έκβαση της διαδικασίας αυτής. Ούτε επίσης τους χρησιμοποιούμε για να αποτιμήσουμε χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Επίσης στηριζόμαστε στην αρχή, στην ε, πραγματική αξία των, ε, ε, των χρηματοπιστωτικών αυτών εργαλείων. Και αυτό ισχύει και για για εισηγμένες στο χρηματιστήριο κεφάλαιο. Η χρήση αυτών των κριτηρίων αναφοράς ελέγχον, ελέγχεται από κανονισμούς. Και η οδηγία, από την οδηγία ΟΣΕΚΑ, ε, καθώς και από τις κατευθυντήρες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής ε, Κινητών Αξιών και Αγορών, που ε, υποχρώνει τα κεφάλαια και τους διαχειριστές να χρησιμοποιούν μόνο αντικειμενικούς δείκτες που πληρούν τα κριτήρια της διαφάνειας σε ό,τι αφορά τις συνιστώσεις και τη στάθμισή τους και επίσης ε, θα πρέπει να είναι με το περιεχόμενο και να έχουν σαφές περιεχόμενο για να μπορεί να ε, υπολογιστεί εκ νέου. Ο κανονισμός για τα κριτήρια αναφορά θα, συ, θα συμπληρώσει και σε μερικά σημεία θα επικαλύψει και τις πρακτικές. Πάντως προϋποθέτει μία στιβαρή επιλογή για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Χάρη διαφάνειας, χάρη διαφάνειας όμως θα ήμασταν υπέρ κάποιων υποχρεώσεων που θα μας επιτρέπουν να λειτουργήσουμε και εμείς σωστά. Ήμασταν ανέκαθεν υπέρ των τριών στόχων της, του κανονισμού της αναλογικότητας σε ό,τι αφορά τα κριτήρια των διαφορών ειδών κριτηρίων αναφοράς με βάση τον κίνδυνο χειραγώγησης. Επίσης της διαφάνειας για να αποφευθεί το κόστος ε, των κριτηρίων αναφοράς που θα μετακυλείται στους ε, τελικούς επενδυτές και επίσης ε, θεμητός ανταγωνισμός για όλους τους δείκτες που, χρησιμοποιούν στην, χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση άσχετα με την προέλευσή τους και να επιτρέπουν την επιλογή μεταξύ μια σειρά έγκυρων, στιβαρών και οικονομικά συμφερόντων κριτηρίων. Η χρήση των ε, benchmarks αυτών θα πρέπει να διακρίνεται από την παραγωγή τους. Επίσης, ε, δείκτες αγοράς που στηρίζονται σε ρυθμισμένα στοιχεία, επίσης θα πρέπει να είναι διαφανείς για τους επενδυτές. Δεν θα επισέλθω σε εξονυχιστικέ λεπτομέρειε γιατί μα τα ανέφερε αυτό ο κύριο Γκραφ. Θα ήθελα να πω ότι ο κανονισμό θα πρέπει να καλύπτει δείκτε που δημοσιεύονται, είναι προσιτέ ε, στο κοινό, γιατί χρειάζεται διαφάνεια για τα στοιχεία των δεδομένων και επίση, ε, πάροχοι τρίτων χωρών δεν θα πρέπει να αποκλείονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα τώρα να διευκρινίσω δύο-τρία από τα σημεία που σα προανέφερα. Καταρχήν για τη χρήση των κριτηρίων αναφορά. Ε, της χρήσης σε σχέση με την παραγωγή των ε, κριτηρίων αναφοράς. Άρθρα 2 και 4. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε τον ορισμό της χρήσης του κριτηρίου αναφοράς για να αποφύγουμε σύγχυση με την ε, θέσπιση του κριτηρίου αναφοράς. Η παρούσα πρόταση δεν ε, εντοπίζει πλήρως όλους τους χρήστες και δημιουργεί προβλήματα στην, στο θεμητό ανταγωνισμό. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στον ορισμό της χρήσης του κριτηρίου αναφοράς με βάση αυτά που συζητά και το Συμβούλιο θα πρέπει ο ορισμός να περιλαμβάνει δύο συγκεκριμένες χρήσεις. Για παράδειγμα, τον συνδυασμό ή τροποποίηση των δικτών σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται νέα στοιχεία, νέα δεδομένα. Επίσης αναφέρεται η χρήση εξωτομικευμένων δικτών από τον διαχειριστή του ενεργητικού. Η αναφορά δικτών που στηρίζονται σε χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφέρθηκε από τον κύριο Γκραφ, γι' αυτό δεν θα επιμείνω σε αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνος χρήση του κριτήριου αναφοράς. Επίσης για την εξέταση της επίδοσης ε, θα πρέπει και αυτό το θέμα να υπαχθεί στις χρήσεις. Γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης ή χειραγώγησης ε, της τιμής εκ μέρους του κεφαλαίου του διαχειριστή. Επιπλέον, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι μόνο δημόσιοι δείκτες ή προσιτοί στο κοινό καλύπτονται. Ο κύριος Γκράφ επισήμανε ότι είναι εκατομμύρια οι δείκτες αυτές. Οι περισσότεροι όμως είναι για θεσμικούς επενδυτές ή είναι αντικείμενο συγκεκριμένης συμφωνίας μεταξύ ε, του επενδυτού και του παρόχου δείκτη. Το άρθρο 3 θα πρέπει να διευκρινιστεί και να αναφέρεται ότι δεν καλύπτονται τέτοιου είδου δείκτε από τον κανονισμό. Επίση, οι επενδυτέ απαιτούν διαφάνεια για τα δεδομένα των κριτηρίων αναφορά και ω προ τη μεθοδολογία, το, τα επίπεδα των τιμών, τη στάθμιση των δικτών σε τακτική βάση. Η διαφάνεια αυτή θα πρέπει να συνδυάζεται και από δηλώσεις για τα κριτήρια αναφοράς και εκεί θα πρέπει να βρίσκουν οι διαχειριστές το κατάλογο με τις υποχρεώσεις που θα πρέπει να πληρώνουν βάσει τις κατευθυντήρες γραμμές και της ΕΣΜΑ. Επίσης θα πρέπει η, διαφάνεια να καλύπτεται και σε μια ιστοσελίδα της ΕΣΜΑ. Αντίστοιχο με αυτό που ισχύει και για τους οίκους αξιολόγησης. Και παραλαμβάνω να μιλούμε μόνο για δείκτες που είναι προσιτοί στο κοινό ή δημοσιευμένοι. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των τρίτων. Συμφωνώ να έχουμε συνθήκε ίσου ανταγωνισμού μεταξύ ε, ενδοκινοτικών και εξοκινοτικών παρόχων. Και μετά από μια μεταβατική περίοδο, που θα είναι τριετής ε, έω πεντετή, θα πρέπει ε, οι ίδιοι οι πάροχοι, αν δεν προβλέπετε κάτι τέτοιο, να αποδεικνύουν την συμμόρφωσή τους με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΙΟΣΚΟ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριο Πιέρ Μάριο Σάτα υπεύθυνο για τα χρηματοοικονομικά της ε, Hypo Bank και μέλος της Unicredit. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ε, κυρίε και κύριοι βουλευτές, μέλη της Επιτροπής σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας αναφέρω κάποιες ιδέες για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα και επίσης να απαντήσω σε ερωτήσεις ενδεχομένως. Η Unicredit ε, καλωσορίζει τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο για τη μεταρρύθμιση της υπάρχουσας δομής και της χρήσης των ευρωπαϊκών κριτηρίων αναφοράς. Νομίζουμε ότι είναι ένα καθοριστικό βήμα για να επανέλθει η αξιοπιστία της αγοράς και να ε, ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη στα κριτήρια αυτά τα πρόσφατα γεγονότα έδειξαν τη σημασία των κριτηρίων αναφορά και πόσο μπορεί αρνητικά να επηρεάσουν του επενδυτέ και του καταναλωτέ ε, λιγότερο προηγμένων χρηματοοικονομικών ε, ε, προϊόντων όπως, όπως οι υποθήκες. Ένα εναρμονισμένο πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιτρέπει να ληφθεί υπόψη και διασυνοριακή διάσταση των κριτηρίων ε, αναφοράς. Θα επικεντρωθώ εδώ στα κριτήρια των χρηματαγορών ε, λόγω της ευρείας χρήσης τους. Ε, η Unicredit έχει χρησιμοποιήσει ένα σύνολο συνεισφερόντων για αυτούς τους καθοριστικούς δείκτες και τα κριτήρια των βασικών χρηματαγορών όπως η Euribor και Όνια και για όλους τους χρήστες των ε, κριτηρίων, καταναλωτές, επενδυτές και όλους τους ε, δημεσάζοντες. Είναι το βασικό στοιχείο οικοδόμησης των χρηματαγορών ε, τα κριτήρια αναφοράς και η έλλειψή τους θα μπορούσε να υποβαθμίσει σοβαρά τις αγορές, να τις πλήξει. Γι' αυτό το λόγο Unicredit θέλει να καταγράφει κριτήρια αναφοράς για τις χρηματαγορές άσχετα από το πρόσθετο κόστος και τις πηγές που μπορεί να, τους πόρους που μπορεί να απαιτήσουν για να δημιουργηθούν αυστηρότεροι κανόνες και να υπάρξει συμμόρφωση. Παρόλο που τα κριτήρια αυτά που ισχύουν σήμερα έχουν δημιουργηθεί πριν από πολλέ δεκαετίε. Βάσει τη πρόταση, η βασική προπόθεση για να θεωρηθεί κρίσιμο ένα δείκτη είναι να έχει υποθετική αξία, υπολογιζόμενη αξία δηλαδή τουλάχιστον 500 δι. Ε, θεωρεί ότι αυτό το μόνο κριτήριο, η Unicredit θεωρεί ότι αυτό το μόνο κριτήριο δεν αρκεί για να θεωρηθεί κρίσιμο ένα δείκτη. Επειδή και κάτω από αυτό το όριο υπάρχει συστημική σημασία των δικτών ε, και των κριτηρίων για πολλά κράτη-μέλη ή για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα ορισμό που να βασίζεται περισσότερο σε ποιοτικά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πρώτα απ' όλα αν χρησιμοποιείται για τη λιανική πώληση και τι χρηματοοικονομικέ συμβάσει, ο δείκτη αυτό, το κριτήριο, ή αν η έλλειψη του κριτηρίου θα μπορούσε να έχει ε, ανεπιθύμητες συστημικές συνέπειες στην χρηματοοικονομική σταθερότητα. Είτε στις αγορές είτε στην πραγματική οικονομία ε, περισσότερων των ενός κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά την εποπτεία θα πρέπει να συμμετέχουν οι αρχές και οι συμβάλλοντες ε, περισσότερο του ενός κράτη μέλη, καθώς και οι χρήστες και η Unicredit θεωρεί ότι η ΕΣΜΑ είναι η ιδανικότερη αρχή για να αναλάβει τέτοιες, αρχές, τέτοιες αρμοδιότητες και εποπτείας. Ο ρόλος της ΕΣΜΑ είναι ζωτική σημασία για τις αποφάσεις ε, που θα αφορούν τους κρίσιμου, τα κρίσιμα κριτήρια αναφοράς και για το γενικό συμφέρον τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χρηματοοικονομικών της ε, αγορών, ε, προκειμένου να αποφευθεί ο κατακαιρματισμός και να κινηθούμε προς μια ένωση των αγορών κεφαλαίων. Τα τελευταία δύο χρόνια περίπου 19 τράπεζες ήρθηκαν από το πάνελ ε, του Euribor. Οι κρίσιμοι δείκτες έχουν λοιπόν διασυνοριακή ε, σημασία και το πάνελ είναι αρκετό, αρκετά μεγάλο, πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο για να εξασφαλίζει την αντιπροσώπευση και την διάρκεια και τη συνέχεια στον χρόνο των ίδιων των κριτηρίων αναφορά. Γι' αυτό το λόγο επίγει να αναλάβει η ΕΣΜΑ αρμοδιότητε ε, που θα επιβάλλουν την υποχρεωτική συνεισφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων και ασχέτω των αριθμητικών ανώτερων ορίων. Βάσει της πρότασης, τα στοιχεία για τις συνελλαγές έχουν προτεραιότητα ως προς την, τον ορισμό των κριτηρίων αναφοράς. Η λογική είναι ότι υπάρχει λιγότερη διακριτική ευχέρεια εδώ και λιγότερη πιθανότητα να είναι αντικείμενο παραποίησης χειραγώγησης στα δεδομένα. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις όπως το μπορεί στα διατραπεζικά έχει εκτιμηθεί ότι μπορεί και αυτά να είναι εύστοχα ε, ε, όταν είναι μεγάλες για τραπεζικές ε, περίοδοι που υπολογίζονται στην αγορά ή όταν δεν υπάρχει αρκετή ρευστότητα και έλλειψη συναλλαγών. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις που να είναι αξιόπιστες και επιτρέπουν να μετρήσουμε την οικονομική πραγματικότητα περίπου σωστά με τα κριτήρια αναφοράς που θα προτιμηθούν. Βάσει της πρότασης οι διαχειριστές πρέπει να δημοσιεύουν τα δεδομένα των συναλλαγών να υπολογίζουν το κριτήριο αναφορά αμέσω μετά τη δημοσίευση του κριτηρίου. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο αν τα δεδομένα αυτά ε, τελικά θα έχουν προστιθέμενη αξία για του χρήστε. Από την άλλη, θεωρούμε ότι η δημοσίευση των δεδομένων των συναλλαγών για τα επιτόκια των αγορών και τα κριτήρια αναφορά του μπορεί να έχουν στρεφλωτικέ συνέπειε σε τράπεζε που θα συμμετέχουν στο πάνελ. Διότι θα αποκαλύπτεται το ε, κόστο χρηματοδότηση των τραπεζών, κάτι που είναι πολύ ευαίσθητο δεδομένο. Ε, έτσι, οι μεμονωμένε τράπεζε και τα επιτόκια του μπορεί να πληγούν μπορούν να ε, πιεστούν και τελικά να υποβαθμιστεί η, συνολική η δυνατότητα της τράπεζας να ε, αντλήσει κονδύλια την αγορά. Οι διαχειριστές λοιπόν πρέπει να, ε, να μην απαιτείται να δημοσιεύουν τα στοιχεία χωρίς κανένα μεσοδιάστημα και μόνον εφόσον το ζητήσει η ΕΣΜΕ εντό ευλόγου χρονικού διαστήματο. Επίση, στον κλάδο εδώ και λίγου μήνε υπάρχουν πρωτοβουλίε για να δούμε κατά πόσον είναι τα κριτήρια αναφορά βιώσιμα, ιδίω για τα επιτόκια αναφορά όπω το Euribor. Ε, Πολλέ από αυτέ τι δυνατότητε είναι ελπιδοφόρε. Ε, τι προοπτικέ είναι ελπιδοφόρε. Όμω, όταν δημιουργήθηκε το Euribor στα τέλη του 1998 περίπου, και εδώ λόγω τη περιπλοκότητα και τη ποικιλία των συμβάσεων που κάλεπτε με διάφορε διαφορετικέ εθνικέ νομοθεσίε, καλό θα ήταν τελικά όλα αυτά να συνοψιστούν σε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία νομοθετική πράξη προκειμένου να μην υπάρξουν διακοπές ή προβλήματα και τριγμοί σε ισχύουσες συμβάσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σάτα. Αυτοί ήταν οι ομιλητές μας. Και τώρα η συζήτησή μας με τα μέλη της Επιτροπής. Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους σε αυτό τον πρώτο γύρο με τον εισηγητή και τους σκιώδης να περιοριστούν στα δύο λεπτά για να ρωτήσουν αυτά που θέλουν. Και παρακαλώ να διευκρινίζετε σε ποιον ομιλητή απευθύνεται το ερώτημα. Και οι ομιλητέ θα έχουν τρία λεπτά για να απαντήσουν. Μετά από αυτόν τον πρώτο γύρο θα έχουμε και μια, ένα γύρο καθιάει. Πρώτος ομιλητής, ο σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚΟ, ο κ. Ντερμάγερ. Δύο λεπτά παρακαλώ για το ερώτηση. Uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να είμαι και πιο σύντομος. Ανησυχώ ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά την, ε, το καθεστώς τρίτου μέρου. Να ρωτήσω του εκπροσώπους τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόβλημα είναι ότι ο κανονισμό καταρτίστηκε κάποια στιγμή που οι αρχέ του ΆΙΣΚΟΚ ε, προετοιμάζονταν. Τώρα λοιπόν έχω την εντύπωση ότι ο ΆΙΣΚΟΚ γίνεται αποδεκτό πλέον ως παγκόσμιο, παγκόσμια αρχή. Άρα σε τι βαθμό είναι ρεαλιστικό να προχωρήσουμε με κάτι που είναι πάνω από τα πρότυπα που ορίζονται από τον Αϊόσκο. Κατά πόσο θα υπάρξει αντίδραση ή κατά πόσο τα άλλα μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα θα προσαρμοστούν στο καθεστώς αυτό. Σε τι βαθμό λοιπόν υπάρχει ο αντίθετος κίνδυνος το δικό μας ε, καθεστώς, η δική μας ρύθμιση να είναι πολύ πιο αυστηρή. Και έτσι να περιορίζονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τη χρήση κριτηρίων αναφοράς εκτός Ευρώπης. Ευχαριστώ και η ερώτηση ήταν προς τον ε, κύριο Επίτροπο, ε, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Φίλιπ Τόντου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να διευκρινίσω το εξής. Το καθεστώς τρατής χώρας έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι τα κριτήρια αναφοράς τρίτων χωρών που χρησιμοποιούνται στα δημοσιονομικά μέσα και στα καταναλωτικά προϊόντα, για παράδειγμα υποθήκες, είναι εξίσου αυστηρά με τα κριτήρια αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και αξιόπιστα. Επίσης, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ίδιους όρους λειτουργίας, όπως και οι ανταγωνιστικές εταιρείες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις πληροδιαγραφές. Είναι σημαντικό το καθεστώς ισοτιμίας μετά την, ε, τον κανονισμό να είναι ε, νομικά σίγουρο για να υπάρχει αυτή η ισότητα. Δεν θεωρούμε ότι η αυτοπιστοποίηση από τρίτες ε, χώρες και από τους πάροχους τέτοιων κριτηρίων αναφορά θα παρέχει ισότητα ευκαιριών και νομική ασφάλεια. Επίσης, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται τόσο πολύ το θέμα των αρχών του ΑΙΟΣΚΟ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη ιδιαίτερως κατά πόσο στο νομικό πλαίσιο των άλλων χωρών και οι υποπτικές τους αρχές εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους ε, κανόνες ΙΟΣΚΟ σε ό,τι αφορά τα benchmarks. Επίσης θεωρούμε ότι η αναθεώρηση του ΙΟΣΚΟ για τη συμμόρφωση της εφαρμογής των αρχών συγγνώμη, θα παράσχει μια χρήσιμη ένδειξη για το κατά πόσον οι χώρες που έχουν προσυπογράψει τις αρχές εφαρμόζουν τις αρχές αυτές και επίσης υπάρχουν διάφορες τρίτες χώρες όπως η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη που εξετάζουν το ενδεχόμενο νομοθεσίας για τα benchmarks με πιο στενό πεδίο εφαρμογής ενδεχομένω αρχικά αλλά με προοπτική διεύρυνση όπως και στο κάτω παρελθόν σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς πιστοποίησης ε, η Ευρώπη ηγείται σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για παγκόσμιες τέτοιε αρχές. Και καλά κάνουμε. Αλλά θεωρούμε από την εμπειρία του παρελθόντος ότι οι τρίτες χώρες ενδεχομένως να ακολουθήσουν και αυτές. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, σκιώδης εισηγητής, ο κύριος Χώνας Φερνάντες. Ευχαριστώ. Συμμερίζομαι και εγώ τον προβληματισμό των συναδέλφων ε, του Έλκαλα. αλλά λάβαμε απάντηση ως προς το ένα σκέλος. Θα ήθελα να, για τον ορισμό του κρίσιμου κριτηρίου αναφοράς να μου πει κάτι εκπρόσωπος της ΕΚΤ. Δεν είναι ιδανικός ο ισχυρός ορισμός. και συμφωνώ ότι η αξιολόγηση των κριτηρίων αναφοράς δεν θα πρέπει να γίνει μόνο με το φως της σταθερότητας της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Μήπως με τον τρέχοντα ορισμό αφήνουμε διακριτική ευχέρεια στις δράσεις του επόπτη. Πώς θα μπορούσαμε να ορίσουμε καλύτερα το κρίσιμο κριτήριο αναφοράς χωρίς να αφήνουμε μεγάλο περιθώριο λιγμό στον επόπτη να αφήνουμε πολλά πράγματα στη διακριτική του ευχέρεια. Επίσης, για τα κριτήρια αναφοράς για τα προϊόντα. Στα κριτήρια αναφοράς για τα προϊόντα, που είναι συνήθως μη χρηματοπιστωτικά κριτήρια αναφοράς, έχουμε πρόβλημα με τους ε, συνεισφέροντες γιατί πολλοί συμβάλλουν ε, με προαιρετικό τρόπο, με εκούσια, σε εκούσια βάση. Στον τρέχοντα κανονισμό έχουμε δεοντολογικό κώδικα που είναι νομικά δεσμευτικός. Και θεωρώ ότι ίσως ε, δημιουργήσει πρόβλημα σε τρίτους που αυτή τη στιγμή σε προαιρετική βάση συμμετέχουν και συμβάλλουν. Πώς θα μπορούσαμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα για τα μη, για τα μη, για τα μη χρηματοπιστωτικά κριτήρια αφοράς και τον κώδικα δεντολογίας που είναι νομικά δεσμευτικός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκιάβη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα του ορισμού του κρίσιμου κριτηρίου αναφοράς λαμβάνονται υπόψη και ποσοτικά και ποσοτικά. Αν ληφθούν υπόψη μάλλον και ποσοτικά και στοιχεία, αναπόφευκτα δημιουργούν και ένα περιθώριο λιγμών και μια διακριτική ευχαίρεια. Αλλά η διακριτική ευχαίρεια προϋποθέτει μια ανάλυση που έχει γίνει από τον αρμόδιο φορέα, από τον φορέα δηλαδή που καταρτίζει αυτή την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης υπάρχει και δυνατότητα αναθεώρησης μετά από κάποιο διάστημα. Οπότε έχουμε μια τελειοποίηση, εξετάζουμε την καταλληλότητα της αξιολόγησης. Είναι σημαντικό όμως να συμπεριληφθούν και τα ποιοτικά και, για τα ποσοτικά στοιχεία. Δηλαδή, αφενός έχουμε εκτεταμένες αναφορές που χρησιμοποιούνται σε πληθώρα συμβάσεων και αφετέρου έχουμε και την ανάγκη της ανάλυσης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που είναι ποιοτικό στοιχείο. Δίνει μια ποιοτική χρειά στην ανάλυση και ισχύει και για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς θέλει το λόγο να απαντήσει στις ερωτήσεις του δεύτερου ομιλητού του. Oh. Δεν είμαι ειδικό ε, περί προϊόντων, αλλά να... μας έχει προβληματίσει και σε σχέση με το Euribor το θέμα αυτό, διότι μέχρι τώρα στηρίζεται σε θελοντική βάση το Euribor. Αλλά με αυτή τη μεταβατική περίοδο υπάρχει μεγάλος κίνδυνος οι τρίτοι συνεισφέροντες να βγουν από το πάνελ. Οπότε τελικά δεν θα δημοσιεύεται ο δείκτη. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει εδώ ο κανόνα τη υποχρεωτική συμβολή βάσει των κανόνων συμπεριφορά. Μάλλον χρειάζεται κάτι αυστηρότερο, Όπω μια νομοθετική πρωτοβουλία και ένα επόπτη που θα επιβάλλει στου συνεισφέροντε στο πάνελ να έχουν υποχρεωτική συμβολή. Επιτροπή, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να απαντήσω στην ερώτηση του βουλευτού για τον κώδικα συμπεριφορά. Να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής σας στις αρχές του ΙΟΣΚΟ που λένε οι διαχειριστές των κριτηρίων αναφοράς να απαιτούν από τους συνεισφέροντος να συμμορφώνονται με τον κώδικα συμπεριφοράς και να την αποδεικνύουν αυτή τη συμμόρφωση ετησίως. Μάλιστα το ίδιο και για όλες τις αλλαγές που θα προκύπτουν στον κώδικα συμπεριφοράς. Έτσι αυτό το κώδικα συμπεριφοράς της ΙΟΣΚΟ ήθελε να αντιγράψει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά πρέπει να εξεύρουμε άλλους τρόπους ώστε η αρχή αυτή να γίνει σεβαστή. Να μεταφερθεί και να γίνει σεβαστή. Η Προεδρία και το Συμβούλιο βρήκαν μια εναλλακτική διατύπωση για να εφαρμοστεί, αλλά αυτήν ακριβώς την αρχή θέλουμε να εφαρμόσουμε εδώ. Ευχαριστούμε για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ο κύριος Σάμπο Τέρχο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματο τη ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, θα ήθελα να κάνω μια γενική ερώτηση προ τον κύριο Ράιτ. Δεν ξέρω αν μπορεί να μα ακούσει. Ναι, κοιτάξτε, λέει ο Πρόεδρο, έχουμε ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη σύνδεση με τη Μαδρίτη. Θα συλλέξουμε τι ερωτήσει για τον Ιώσκο στο τέλος. Α, έχω άλλη μια ερώτηση να κάνετε, βεβαίω. Ναι. Να θέσετε τη δεύτερη ερώτησή σα. Ναι, και πιο συγκεκριμένη ερώτηση για τον κύριο Γκράφ. Κύριε Γκράφ, ε, ω εκπρόσωπο τρίτη, ε, χειριστή μάλλον ε, εκπροσώπου τρίτη χώρα για τα κριτήρια αναφορά. Τι γίνεται με το ίδιο πεδίο εφαρμογή, υπάρχουν τέτοιες προ... υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό, όπω και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, η ελβετική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη, δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματής Έχουν γίνει διάφορες αρχικές συζητήσεις και ως τώρα δεν υπάρχει προετοιμασία νομοσχεδίου. Δεν υπάρχει σχέδιο εφαρμογής νομοθεσίας για τους δείκτες στην Ελβετία. Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε στο ερώτημά σας όταν θα είμαστε και πάλι σε σύνδεση με τον Ιώσκο. Ο κύριος Βίγκας. Euh, Καταλαβαίνουμε τη σημασία αυτών των κριτηρίων αφορά και μα το δείχνουν και οι εμπειρίε του πρόσφατου παρελθόντο. Τεράστιε ζημιέ που έχουν προκύψει από την ε, παραποίηση τέτοιων ε, δικτών όπω συμβάσει SWAP ε, με κρατικές επιχειρήσεις και με, εξωτερικό, με εξωτερικές δαπάνες δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά όλα επιβεβαιώνουν όσο υπόθηκαν. Οπότε αυτές οι ατασταλίες, αυτές οι καταχρήσεις προκύπτουν από την συμβολή δύο παραγόντων. Πρώτα απ' όλα σύγκρουση συμφερόντων, όπου μετά ε, και η υπερπλοκότητα των δικτών έρχονται να επιβαρύνουν τα πράγματα. Δηλαδή, ο τρόπος που δομούνται τα κριτήρια αυτοί προκαλούν και προξενούν αυτά τα προβλήματα. Σε αυτό το υποθέτη διάσταση καλό θα ήταν να φροντίσουμε για την καλή ποιότητα και το εύληπτο αυτών των κριτηρίων αναφοράς εφόσον είναι κάτι τέτοιο εφικτό. Η ερώτηση που ήθελα να θέσω στους διάφορους ομιλητές είναι μήπως ήταν ευστοχότερο σε αυτό το πλαίσιο να δώσουμε ένα σημαντικότερο ρόλο στις ε, δημόσιες παρεμβάσεις. Δηλαδή στις δημόσιες αρχές έχουμε ε, αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη που θα μπορούσαν να έχουν πολύ καθοριστικότερο ρόλο να διαδραματίσουν στο θέμα αυτό. Αυτό θα ήταν μια σωστή κίνηση εφόσον θεωρούμε ότι αυτά τα κριτήρια αναφοράς που έχουν τέτοια οικομενική χρήση παντού ε, έχουν και δημόσια αξία, ε, είναι δημοσίου συμφέροντος. Σε ορισμένα λοιπόν από τα κριτήρια αναφοράς, γιατί μια, αρχή όπως η Eurostat, η, η EFA να μην αναλάβουν τον καθορισμό ενός κριτήριου αναφοράς και εφόσον ίσως να προλαμβάνει τις συγκρούσεις συμφερόντων κατά αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε. Θέλετε να απαντήσετε. Μάλλον θέλετε να ρωτήσετε κάποιον συγκεκριμένο ή να απαντήσουν όλοι. Ποιος θα ήθελε να απαντήσει. Τι δημόσιο ρόλο θα μπορούσαμε να προβλέψουμε για συγκεκριμένα κριτήρια. Παρακαλώ, Κεντρική Τράπεζα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Βουλευτά. Ο δημοσίος τομέας νομίζω ήδη έχει κάνει πολλά. Ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα οι επόπτες δεν είμαστε εμείς αυτή την περίοδο που αναφέρεται. Πριν από δύο μέρες περίπου αναλάβαμε. Αλλά τέλος πάντων τώρα έχουμε και εποπτικές αρμοδιότητες. Και έχουμε αρμοδιότητα για την προληπτική διάσταση και όχι για την ε, διεξαγωγή των χρηματοοικονομικών ε, δραστηριοτήτων. η εποπτεία ήταν διαφορετική όταν προέκυψαν αυτά τα σκάνδαλα και όλε αυτέ τι παραποίησει. Επίση, οι κεντρικές, η κεντρική τράπεζα από την πλευρά τη συμμετείχε ενεργά προκειμένου να στηρίξει τι διαδικασίε μεταρρύθμιση. Όλοι οι ομιλητέ σχολίασαν το τι γίνεται με τις διάφορες εκθέσει και τι ομάδε που υπό την αιγίδα του BIS, του ΑΙΟΣΚΟ και του Συμβουλίου για την Χρηματοοικονομική Σταθερότητα ασχολήθηκαν με, τα, με τις ισοτιμίες αναφοράς. το μήνυμα της ακεραιότητας έχει γίνει αντιληπτό ακεραιότητα και στην ε, συμπεριφορά των ε, συνεισφερόντων αλλά και στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για να υπολογιστούν τα κριτήρια αναφοράς. Στο μήνυμα αυτό επιμένουμε έκτοτε με την ενεργό μας συμμετοχή ε, ως ε, έχοντας καταλητικό ρόλο για την μεταρρύθμιση των πρωτοβουλειών των δρόντων στην αγορά, των διαχειριστών του Euribor. του να δημιουργηθεί ένα Euribor αναφοράς που να βασίζεται στις συναλλαγές λόγου χάρη. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Να προσθέσω μία σύντομη πληροφορία. Φυσικά και ο ιδιωτικός κλάδος καταβάλει προσπάθειες για, να, για αποκατάσταση της διαφάνειας των κριτηρίων αναφοράς των benchmarks και προσπαθεί να αποκαταστήσει τη μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτή την αγορά που στηρίζεται περισσότερο σε υποκειμενικά κριτήρια, να στηρίζεται σε κριτήρια συναλλαγής. και αν εξωθήσουμε ε, τον ιδιωτικό κλάδο εκτός περιεφαρμογής ε, θα περιορίσουμε τις δυνατότητες ε, σχεδιασμού και θέσπισης κριτήριων αφοράς με βάση τα κριτήρια της συναλλαγής. Επαναλαμβάνω ότι και για αυτό το τμήμα καταβάλει μεγάλη προσπάθεια ο ιδιωτικός κλάδος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φίλιπ Λάμπερτς από τους ε, Πρασίνους. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς θα προτιμούσαμε να καλύπτονται όλοι οι δείκτες από τον κανονισμό. Με διπλή προσέγγιση όμως τα μη κρίσιμα κριτήρια αναφορά να υπόκειται σε ένα πιο light καθεστώ και τα κρίσιμα στοιχεία αναφορά να υπόκειται σε ένα πιο αυστηρό καθεστώ. Αλλά να καλύπτουμε όλα τα κριτήρια αναφορά, όλου του δείκτε. Και αν ε, ένα κριτήριο αναφορά περάσει από την μη κρίσιμη στην κρίσιμη κατηγορία να καλύπτεται ανα πάσα στιγμή και να υπόκειται σε εποπτεία. Ποια είναι η, η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την πρόταση αυτή. Και έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φαίνεται ότι δημιουργήθηκε περιττός κίνδυνο στι χρηματοπιστωτικές αγορές από το γεγονός ότι τα κριτήρια αναφοράς χρησιμοποιούνται για κατάλληλε συναλλαγέ. Το LIBOR χρησιμοποιήθηκε σχεδόν για τα πάντα αυτό το διατραπεζικό επιτόκιο του Λονδίνου, ακόμη και όταν ήταν άσχετο με τη χρήση. Πώ μπορούμε λοιπόν, ερωτώ, να αντιμετωπίσουμε αυτή την ακατάλληλη χρήση των κριτηρίων αναφοράς, πώς να προβλέψουμε νομοθετικές διατάξεις για να αποφύγουμε τέτοια ανάρμοστη χρήση, ώστε να χρησιμοποιούνται αυτά τα κριτήρια να αναφορά μόνο όπου δει και όχι με ακατάλληλο τρόπο, γιατί αν, χρησιμοποιηθεί, αν χρησιμοποιηθούν με ακατάλληλο τρόπο για ανάρμοστες ε, συναλλαγές θα πρέπει να εντοπίζουμε τον κίνδυνο και να, επικεντρώνουμε την προσοχή μας αυτό. Κύριε Γκραφτ. Ε, έχετε κάποια ιδέα για το εύρος ε, της χειραγώγησης που γίνεται σε τέτοιου είδους ε, δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για να απαντήσω στην ερώτηση για το πώς να καλυφθούν διάφορες, διάφοροι δείκτες και ίσως κάποιοι δείκτες να υπόκεινται σε πιο σε λιγότερο αυστηρό καθεστώ, θεωρούμε ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό ακριβώ κάνει. Δεν λέμε ότι είναι τέλεια και σαφώ και υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέχει κάποιε οριζόντιε κοινέ ε, αρχέ και απαιτήσει για όλου τα κτίρια αναφορά και προβλέπει πιο αυστηρά κριτήρια για τα κρίσιμα κριτήρια αναφορά σε υπερβολικές, χρεωτικέ ε, συνεισφορέ και σε ό,τι αφορά την αναγνώριση από άλλους, από τρίτα μέρη, από τρίτες χώρες και συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους ρυθμισμένα κριτήρια απόφασης δεδομένων όπου προβλέπουμε απαιτήσει που προβλέπονται και σε άλλα σημεία της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες ε, προδιαγραφές για τα benchmark των ε, με επιτόκια και συγκεκριμένων εμπορευμάτων. Προβλέπονται λοιπόν ειδικά καθεστώτα για κάποια είδη benchmarks, αλλά θεωρούμε ότι όλα τα κριτήρια αναφοράς θα πρέπει να ρυθμίζονται δημόσια και να βρίσκονται υπό δημόσια υποπτία, γιατί θεωρούμε ότι όλα τα benchmark υπόκεινται σε παρόμοιους κινδύνους. Δεν θα θέλαμε λοιπόν και να παραθυράκια στην νομοθεσία μας, τα οποία στο μέλλον ενδεχομένως να εμφανιστούν όταν θα εμφανιστούν και νέα σκάνδαλα στην χειραγώγηση κριτηρίων αναφοράς. Βλέπουμε ότι διάφορα σκάνδαλα πάνε και πολύ παραπέρα από τα κριτηρία αναφοράς. Είδαμε ότι υπήρξαν αιτιάσεις χειραγωγάγησης σε ό,τι αφορά ε, κριτήρια αναφοράς, ε, εξωτερικού συναλλάγματος, ε, εμπορευμάτων. Καλό λοιπόν να υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο για όλα τα κριτήρια αναφοράς και βλέπουμε μετά πώς θα είναι πιο προσαρμοσμένα από τα δευτερεύοντα κριτήρια, τα δευτερεύουσε προδιαγραφέ όπου υπάρχουν συγκεκριμένε ανάγκε. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τώρα, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άξιο ότι είμαι οι βουλευτέ. Εγώ θα έλεγα το εξή. Από την αρχή του 2013, εμείς ως κεντρική τράπεζα υπό την αιγίδα του EBIS. Δημοσιεύσα, δημοσιεύσαμε μία έκθεση που περιλαμβάνεται και δημοσιεύτηκε και στην ιστοσελίδα της τράπεζας. Ιδιαίτερος αναφέραμε την αρχή της επιλογής. Αυτό ακριβώς νομίζω υπονοούσατε και σας ευχαριστώ που το θέσατε αυτό ως θέμα. Μας απασχολεί ιδιαίτερως η αρχή λοιπόν του να επιτρέψουμε στους συμμετέχοντες της αγοράς, στους οικονομικούς φορείς και στους τελικούς χρήστες να επιλέξουν μεταξύ των διαφόρων δικτών, των διαφόρων κριτηρίων αναφοράς προκειμένου να βρουν τι ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους. Γι' αυτό λοιπόν τονίσαμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ποικιλία και ότι πόσο σημαντική είναι για την ανάλυση στο τέλος ο τελικός χρήστης να μπορεί να συνδέσει τις διάφορες επιλογές του με την ανάγκη και με τη χρήση ενός κάποιου κριτηρίου αναφοράς. Σωστά επισημάνατε και αναφέρετε ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα κριτήρια αναφοράς, για παράδειγμα, των συναλλαγματικών ισοτιμιών των επιτοκίων περιλαμβάνουν τον ε, βάθμο κινδύνου και όλα αυτά που περιλαμβάνονται στις αναφορές τους και ότι αυτά χρειάζονται για να ε, καθοριστούν τελικά σε συγκεκριμένες επαφές. Αυτή η φιλοσοφία δε μπαίνει και στην προσέγγιση του της Επιτροπής ε, Οικονομικής Σταθερότητας, όπου αναφέρεται ότι υπάρχει μια Εποπτική Επιτροπή και σε αυτήν συμμετέχουν και οι κεντρικές τράπεζες προκειμένου να βοηθηθούν οι φορείς της αγοράς για να βρουν μια προσέγγιση διαφόρων τιμών για την Ευρωζώνη για παράδειγμα. Ήδη έχουμε κάτι που είναι που είναι ένα επιτόκιο χωρίς σχεδόν κίνδυνο και μια τιμή όπως το Euricor που περιλαμβάνει τον κίνδυνο αυτό. Είναι νομίζω ύψης της σημασίας να διασφαλίσουμε την σταθερότητα και την συνέχεια τέτοιων κριτηρίων αναφοράς. Τώρα, πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά να τον αποφύγουμε ακατάλληλα στοιχεία, την προστασία των ε, πελατών. Όπως σας είπα, νομίζω πιο αρμόδιος θα ήταν ε, για να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι η Κεντρική Τράπεζα. Αλλά κάνουμε κάτι απτό. Δημιουργούμε μία ποικιλομορφία, την επιλογή. Τα υπόλοιπα, θεωρώ, θα πρέπει να τα αφήσουμε στα χέρια των ε, οργάνων που είναι υπεύθυνα για την προστασία. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε παρακαλώ να ακούσουμε και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σημείο αυτό. Ναι, το συγγνώμη που παρέλειψε τη δεύτερη σας ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί μαζί σας ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε και αυτό το θέμα. Δηλαδή το θέμα της καταλληλότητας των κριτηρίων αναφοράς που θα πρέπει να αξιολογείται ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται σε χρηματοπιστωτικές συμβάσει με καταναλωτέ, Γι' αυτό και το, έχουμε το άρθρο 18 για την αξιολόγηση της καταλληλότητα, που λέει ότι πριν την υπογραφή χρηματοπιστωτικής σύμβασης με καταναλωτή που παραπέμπει σε κριτήριο αναφοράς, η εποπτική αρχή θα πρέπει να ελέγξει την πείρα και γνώση του καταναλωτή ό,τι αφορά το κριτήριο αναφοράς, την οικονομική του κατάσταση και τους στόχους και να κρίνει κατά πόσο αυτό το κριτήριο αναφοράς είναι κατάλληλο για τον συγκεκριμένο καταναλωτή, για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Και αν μετά από αξιολόγηση η εποπτική αρχή θεωρήσει ότι το κριτήριο αναφοράς είναι κατάλληλο, θα πρέπει γραπτός και αιτιολογημένο να ενημερώσει τον καταναλωτή, ώστε να αποφασίσει αν θα υπογράψει τη σύμβαση ή όχι, αν θεωρήσει ότι είναι ακατάλληλο το κριτήριο αναφοράς για αυτόν. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και φροντίσαμε να το καλύψουμε στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Και τώρα έχει το λόγο και πάλι η συγγετριά μας, η Κόρα Βαν Ιβενχόιζεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλές είναι οι ερωτήσεις που ήδη τέθηκαν και απαντήθηκαν. Εγώ να επανέλθω σε μια ερώτηση που την έθεσε και ο κύριος Φερνάντες για την ε, κρισιμότητα κάποιων κριτήριων αναφοράς. Ο κύριος Σκιάβη και ο κύριος Σάτα επειδή και οι δύο εκφράστηκαν ε, για τους ορισμούς των κρίσιμων ε, δικτών και το ποιοτικό, το ποσοτικό μάλλον όριο που προβλέπετε και το τι γίνεται με την υπέρβαση του όριου αυτού από κάποια κριτήρια αναφοράς. Είπατε κύριε Σκιάδη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει έναν πιο ευέλικτο, ε, περισσότερο διαλεκτικό ορισμό για τον ορισμό των κρίσιμων κριτηρίων αναφορά. Πώ το βλέπετε δηλαδή αυτό το ποσοτικό όριο τελικά και ε, πιο συγκεκριμένα τι ποιοτικά κριτήρια θα θέλατε να χρησιμοποιηθούν για τον ορισμό των δικτών. Διότι λέτε ότι θα πρέπει τα επιτόκια να τα ε, αν, κοιτάζουμε από καιρού εις καιρών και οι αρμόδιες αρχές να κάνουν τις κατάλληλες ε, αποτιμήσεις. Ποια είναι η άποψή σα και το ίδιο ρωτώ και τον κύριο Σάτα. Και αν με επιτρέπετε, Πρόεδρε, θέλω και άλλη μια τελική ερώτηση προ τον κύριο Σίμπελ. Ε, είπατε ότι τα επιτόκια χρησιμοποιούνται για να μετρηθούν οι επιδόσεις των επενδυτικών ε, ταμείων, αλλά δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο αυτού του κανονισμού. Γιατί δεν θα προκύψουν προβλήματα σύγκρουσης συμφερόντων και ε, προσπάθειες παραποίησης σε ό,τι αφορά τέτοια, αυτά τα κριτήρια αναφοράς. Τι σας κάνει να το πιστεύετε. Πρόεδρος. Ποιος θέλει. Κύριε Σάτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο λόγος για τον οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ένα όριο δεν είναι ίσως ο καταλληλότερος είναι ότι κάποιες από τις χρηματαγορές που έχουμε υπόψη και στις οποίες αναφέρονται τα κατήρια αναφοράς είναι αγορές πολύ δύσκολο να μετρηθούν ως προς τον ακριβή τους όγκο ή τις αναλογίες που λαμβάνουν χώρα εκεί. όχι μόνο για τα εργαλεία που συνδέονται αμέσω απευθεία με τα κριτήρια αναφορά, αλλά και πολλά από αυτά που συνδέονται με τα μόχλευση. Οπότε, οι πάροχοι των ε, ε, κριτηρίων αναφοράς μπορούν οι ίδιοι να παρακάμψουν ε, τα τα όρια. Ενώ αν οι αρχές χρησιμοποιούσαν ποιοτικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με το εύστοχο των δικτών, θα ήταν πολύ καλύτερα. Ένα παράδειγμα. Δεν μιλάμε μόνο για το συνολικό όγκο ε, που χρησιμοποιείται ως βάση υπολογισμού για τα κριτήρια αναφορά, αλλά και για τη σημασία των δικτών. Το Euribor είναι σημαντικός, σημαντικό επιτόκιο, όχι μόνο γιατί είναι τεράστιος όγκος των συναλλαγών που αφορά, αλλά γιατί αφορά και ε, υποθήκες λιανικής και για όλους αυτούς τους λόγους είναι μεγάλη σημασία του. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο η αριθμητική προσέγγιση η ποσοτική προσέγγιση. Ε, με έναν ακριβή ορισμό περί ποιοτικής προσέγγισης θα ήταν καλύτερο και για σκοπούς χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Και αυτό θα πρέπει να το αποφασίσουν οι ε, επόπτες. Είναι ε, ένα συμβιβασμό αυτός φυσικά, γιατί η διακριτική ευχέρεια δεν θα καταργηθεί, αλλά νομίζουμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να καλύψουμε το θέμα αυτό. Κύριε Σκιάβη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Συγήτρια. Προσπαθούμε να ποσοτικοποιήσουμε ποιοτικά στοιχεία. Βέβαια, αυτό είναι μια μεροληπτική στάση οικονομολόγου ίσως. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Σάτα και κάποια άλλα μέτρα. Για παράδειγμα, λαμβάνουμε υπόψη, αξιολογούμε τη σημασία ενός δίκτυ για συγκεκριμένη χώρα. Δηλαδή, ποιο είναι το μέγεθος των οικονομικών, της οικονομικής δραστηριότητας ε, ή όγκος των συμβάσεων σε μια συγκεκριμένη χώρα που σχετίζονται με συγκεκριμένο δίκτυο και ακόμη και αν ο ε, λόγο δείκτης μπορεί να μην χρησιμοποιείται ευρέως, ίσως σε μια χώρα δημιουργήσει πρόβλημα ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα που μπορεί στη συνέχεια να μεταδοθεί και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, θα πρέπει να δούμε και το είδο των συμβάσεων ε, για τι οποίε χρησιμοποιούνται τα κριτήρια αναφορά. Για παράδειγμα, θα πρέπει να δούμε κάποια Μία χρησιμοποιείται ή κάποια αναφορά χρησιμοποιείται από πιο επαγγελματικά ιδρύματα ή υπηρεσίες ε, ή ποιοι είναι οι τελικοί χρήστες, μήπως είναι απλοί καταναλωτές. Οπότε η σύνδεση της ε, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του συστήματος ε, πώς συνδυάζεται με συγκεκριμένη αναφορά. Συμφωνώ με τον κύριο Σάτα τέτοιου είδους ε, συμπληρωματικοί δείκτες βέβαια θα προσφέρουν και ένα ποιοτικό στοιχείο στην αξιολόγηση για ένα κατώτατο όριο που θα ισχύει για όλους. Και αν ε, πέσουμε κάτω από το κατόφλι της κρισιμότητας, ε, το το πλαίσιο δεν είναι τόσο αυστηρό. Ευχαριστώ κύριο Ζίμπελ. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα έλεγα ότι δεν υπάρχει καθόλου σύγκρουση αλλά ε, είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες. Και οι εταιρείε ε, διαχείρισης ε, κονδυλίων χρησιμοποιούν, διαχειρίζονται 13 εκατομμύρια ευρώ. Και ένα μεγάλο τμήμα είναι ο ΣΕΚΑ. Και χρησιμοποιούν κριτήρια αναφορά για να αποτιμήσουν τις δικές τους αποδόσεις. Και όλα, όλοι οι ΟΣΕΚΑ, όπως ξέρετε, επιβλέπονται από τις εθνικές αρχές με συντονισμό της ΕΣΜΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών. Και η οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ και η οδηγία για τα επιλέξιμα στοιχεία του ενεργητικού, αλλά και οι τελευταίες κατευθυντήρες γραμμές ε, για τα εισηγμένα στο χρηματιστήριο κεφάλαια προβλέπουν πολλές, ε, πολλά πολλές απαιτήσει για την καταλληλότητα και για τη διαφάνεια. Οπότε η ρυθμιστική αρχή έχει και το χρόνο και τις πληροφορίες ε, να ζητήσει από τον διαχειριστή των στοιχείων του ενεργητικού στοιχεία ώστε να δει αν το κριτήριο αναφοράς που χρησιμοποιείται, που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη απόδοση. Για παράδειγμα, για ίδια κεφάλαια χρησιμοποιείται, αν μιλούμε για διαχείριση ιδίων κεφαλαίων αμοιβαίων. Επίσης, ε, είπαμε ότι δεν επηρεάζουμε άμεσα την αποτίμηση της τιμής ενός προϊόντος. Και οι ΟΣΕΚΑ αγοράζουν ε, ε, προϊόντα και κεφάλαια που στηρίζονται σε ρυθμισμένες τιμές και λαμβάνουν υπόψη την καθαρή αξία. Επίσης, η σύγκρουση συμφερόντων είναι περιορισμένη γιατί χρησιμοποιούμε δείκτες και κριτήρια αναφοράς ε, που είναι κρίσιμα ή ρυθμισμένα και τα περισσότερα, τις περισσότερες φορές οι δείκτες στηρίζονται σε ρυθμισμένα δεδομένα. Οπότε αυτή την άποψη δεν μπορεί να δημιουργηθεί σύγκρουση συμφερόντων. Πάντως, ο συνδυασμός της καταλληλότητας του δείκτη που ελέγχεται και απαναθεωρείται από τον ρυθμιστή των κεφαλαίων αλλά και η αξιολόγηση που γίνεται περιορίζει το ελάχιστο τη σύγκρουση συμφερόντων. και η χρήση των ε, ρυθμισμένων δικτών για την αποτίμηση της απόδοσης ε, θα πρέπει να θεωρείται τελική χρήση και όχι παροχή. Γι' αυτό και θα πρέπει να αποκλείεται από την πρόταση του Συμβουλίου. Ευχαριστώ και φαίνεται ότι τώρα έχουμε πλέον σύνδεση με τη Μαδρίτη. Σωστά να δώσουμε το λόγο στον ε, κύριο Τέρο για να θέσει την ερώτησή του λοιπόν. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ελπίζω να μας ακούτε κύριε Ράιτ. Σας παρακαλώ, πείτε μας τι άλλες δικαιοδοσίες εντός της ΙΟΣΚΟ σκοπεύουν να εισαγάγουν συγκεκριμένη νομοθεσία για τα κριτήρια αναφορά που θα καλύπτουν το ίδιο πεδίο εφαρμογή όπως και το σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύετε επίσης ότι οποιαδήποτε δικαιοδοσία στον κόσμο θα μπορούσε να καλύπτει και να πληρεί τους όρους για τις τρίτες χώρες όπως ε, προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο κανονισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ράιτ έχει το λόγο. Mr. Wright. you can, Αν θέλετε να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και πολύ λυπάμαι που υπάρχει δυσκολία και δεν μπορώ να παρακολουθήσω τη σημαντική συζήτηση. Να απαντήσω την τελευταία ερώτηση πρώτα. Με ακούτε? Ναι, σας ακούω, αλλά δεν με ακούτε εσείς. Ναι, σας ακούμε. I can hear you. Hmm? Yes, you can, you can answer. Okay. You can talk. It's okay for us. Have difficulty hearing uh, all the uh, important debate. Okay, let me continue. Να συνεχίσω λοιπόν. Για την ερώτηση σχετικά με τις άλλες ε, δικαιοδοσίες, κατά πόσον σχεδιάζεται ε, νομοθεσία Εξ όσων γνωρίζουμε, μόνο η Ιαπωνία και το Χονγκ Κόνγκ, αλλά με πολύ στενό πεδίο εφαρμογής προγραμματίζουν να περάσουν νομοθετικά μέτρα. Και νομίζω ότι όντως ε, αληθεύει ότι καμία δικαιοδοσία, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν πρόκειται να φτάσει εκεί που έχει φτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο κανονισμού της και στις διαπραγματεύσεις της. Ε, Ακούσαμε κάτι για το καθεστώς ε, τρίτων χωρών, αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητά μέλη. Θα ήθελα να πω το εξής. Έχουμε ένα παράδειγμα με τα παράγωγα στην παρούσα φάση, όπου η ΕΠΑ ενέκριναν κανόνες για τα παράγωγα πολύ, πάνω, πολύ πριν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έκτοτε προσπαθούμε να συνενώσουμε δύο συστήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουμε αυτό. Ως εκ τούτου, αυτό που θέλω να πω στην παρούσα φάση είναι ότι θα ήταν ιδανικά τα πράγματα αν αποτελούσαν τη βάση αναγνώρισης των ε, κριτηρίων αναφοράς οι κανόνες του ΙΟΣΚΟ και θεωρώ ότι τώρα είναι η στιγμή. Προτού εμφανιστούν τα προβλήματα σε διασυνοριακό επίπεδο όσο πιο δυνατό, όποιο γρήγορα δυνατόν μπορούν να ξεκινήσουν οι συζητήσεις, τόσο το καλύτερο. Ο αξιότιμος κ. Λάμπερτ ε, σχολίασε τη χρήση των ε, κριτηρίων αναφοράς και νομίζω ότι έθεσε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο όντως συμπεριλαμβάνεται στο έργο για την ε, χρηματοοικονομική σταθερότητα και για την φάση μετάβασης. Η FSB προτείνει μια διτή προσέγγιση όπου αναφέρεται ο κίνδυνος ε, για τα τραπεζικά δάνεια και προτείνεται το σύστημα IMO+. Όπου χρειάζονται όμως ε, τιμές ε, χωρίς κίνδυνο, προτείνεται εναλλακτική προσέγγιση. Και προφανώς το δύσκολο είναι οι μεταβατικές ρυθμίσεις. Ο κ. Λάμπερτς ρώτησε για την έκταση της χειραγώγησης. Δεν μπορώ να δώσω συγκεκριμένη απάντηση περίπου 5-3 εκατομμύρια δολάρια α, κάθε ημέρα περιλαμβάνει αυτή η αγορά. Όλοι λοιπόν γνωρίζουν τις διάφορες έρευνες που γίνονται για τη χειραγώγηση της αγοράς αυτής και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όπως και όλοι σας διαβάζω εφημερίδες και βλέπουμε ότι διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν προβλέψει σημαντικά ποσά για μελλοντικά ενδεχόμενα πρόστιμα. Θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν την έκβαση των, μελετών, των ερευνών αυτών. Ευχαριστώ. And... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ράιτ. Ελπίζουμε να είναι καλύτερη σύνδεση την επόμενη φορά. Okay. So now we have some time. Τώρα έχουμε λίγο χρόνο για ένα γρήγορο catch the eye. Υπάρχει κάποιος που θα θέλει το λόγο για να θέσει ερώτηση προς τους προσκεκλημένους μας. Μάλιστα. Η κυρία Ντότζ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Ο καθένας από τους ομιλητές είπαν ότι συμφωνούμε το πνεύμα αυτής της νομοθετικής πρότασης. Όμως, για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση, πρέπει να συμφωνήσουμε και στην πράξη με το πνεύμα αυτό. Έγινε πολλής λόγος για το πώς θα βεβαιωθούμε ότι τα διάφορα στοιχεία της ε, νομοθεσίας θα είναι αρκετά συνοσφαιρικά και αξιόπιστα. Νομίζω ότι κάτι που μας λείπει από την αρχή στην ε, θεώρηση του όλου θέματος. Είναι ένα θέμα νοοτροπίας. Οι πελάτες έχουν την εντύπωση ότι δεν την κάνουν δικής μεταχείρισης. Αυτό είναι θέμα νοτροπίας και ψυχολογίας. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν και κανόνες δικαιοσύνης για τη συμπεριφορά προς τους πελάτες. Ε, η ερώτησή μου λοιπόν είναι μάλλον προς τον κύριο Σάτα που το ανέφερε. Αισθάνεται ότι η νομοθεσία που προτείνεται έχει να κάνει με το πώς γίνεται αντιληπτή η συμμόρφωση. Ε, δηλαδή θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει προθεμία να φερθεί κανείς δίκαια στους πελάτες του, μήπως αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Κύριε Σάτα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί είναι σημαντικό όταν μιλάμε για τα κριτήρια αναφορέ, να διακρίνουμε δύο σημαντικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα ο σχεδιασμός των δικτών και μετά τι είδου χειραγώγηση έχει συμβεί. Η χειραγώγηση είναι αδίκημα, έχει συμβεί και πρέπει να διωχθεί. Εδώ, όταν μιλάμε στο επίπεδο του σχεδιασμού, η νομοθετική αυτή πράξη είναι πολύ καλή και πολλές φορές μπερδεύουμε και τα δύο, γιατί μιλάμε για δεδομένα βάση των συναλλαγών. Αυτό μπορεί να βοηθήσει για να αποφύγουμε την παραποίηση της παραπιάσης. Αλλά όχι πάντοτε στις, στις αγορές χωρίς ρευστά προϊόντα. Δεν είναι τόσο σημαντικές. Η νομοθεσία λοιπόν πρέπει να καλύπτει και τα δύο σκέλη. Και το σχεδιασμό, καθώς προσπαθούμε να κινηθούμε προς κριτήρια αναφορά που να είναι τακτικά στην χραγωγήση, αλλά δεν μπορεί να είναι και τελείω προστατευμένα. Οπότε θα πρέπει να ισχύουν κάποιοι κανόνε χρηστή διακυβέρνηση και νομίζω ότι το σχέδιο αυτοκανονισμού είναι πολύ καλό για τη διακυβέρνηση και τον έλεγχο. Εφόσον είναι εφαρμοστεί, θα βοηθήσει πολύ. θα βοηθήσει και στο επίπεδο των συμβαλόντων και των όσων υπολογίζουν. Τα κριτήρια Ναι, μόνο μία σημείωση. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Πιστεύουμε ότι οι χρήστες επίσης έχουν καλύτερη ψυχολογία πλέον και καλύτερη νοοτροπία εμείς ως χρήστες και εσείς στο Κοινοβούλιο κάποιες φορές έχουμε εκπλαγεί με τα πώς έχουν τύχει χειραγώγησης κάποια από, τα, κάποια από τους δείκτες των χρηματαγορών. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι Ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση προς τον κύριο David Ράιτ της Ιόσκο. Είπατε ότι μόνο η Ιαπωνία και το Χονγκ Κόνγκ εξετάζουν νομοσχέδια για το θέμα αυτό. Βέβαια και οι δικές σου νομοθετικές διατάξεις δεν θα είναι τόσο απαιτητικέ. Θεωρείτε ότι είναι δυνατό η ενωσιακή νομοθεσία να προκαλέσει ε, ανταγωνιστικό μειονέκτημα ή ε, να πλήξει την ανταγωνιστικότητα των εταιριών που χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά κριτήρια αναφορά σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο που δεν τα χρησιμοποιεί. Μήπως καλό θα ήταν να έχουμε ενιαίο κανονισμό ώστε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παντού να δρούμε το, ε, με τον ίδιο τρόπο και να έχουμε παγκόσμια κριτήρια αναφορά. Γιατί αυτή η περίπτωση δεν θα χρειαζόμασταν ευρωπαϊκά κριτήρια αναφορά. Νομίζω ότι μόνο παγκόσμια κριτήρια αναφορά θα εξασφάλιζαν συνθήκε θεμητού ανταγωνισμού παντού στον κόσμο. Ευχαριστώ. Κύριε Ράιτ, παρακαλώ. Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα με τον ήχο. Υπάρχουν πολλές παρεμβολέ. Yeah, Mr. Wright, Do you, yes, please. That's a very um, interesting thought uh, from the honorable. Ενδιαφέρουσα η σκέψη σας. Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν πρόκειται να έχουμε ενιαία κανονιστική διάταξη, ενιαίες ρυθμίσεις. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συζητούμε όλο και περισσότερο για να συγκλίνουμε κάπως απόψεις μας. Τίποτα όμως δεν είναι νομικά δεσμευτικό. Ούτε ό,τι κάνουμε εμείς, ούτε η Συμφωνία Βασιλεία, ούτε άλλες ε, διεθνείς συμφωνίες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει στο εγγύς μέλλον. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Υπάρχουν κάποιες αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο και ελπίζουμε να εφαρμόζονται γενικώ όπου χρειάζεται. Και αυτό είναι μια απόφαση που θα λάβει κάθε δικαιοδοσία από μόνη της.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 Thank you Σας ευχαριστούμε, κύριε Ράιτ. Δεν ζητά άλλος κανείς το λόγο, οπότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και τη δημόσια κρόση, δίνοντας και πάλι το λόγο στην εισηγητριά μας, την Κόρα. Θα είμαι λακωνικότατη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας και όλους όσους έλαβαν μέρος ε, στην δημόσια αυτή ακρόση, ιδιαίτερα τους εμπειρογνώμονές μας, ε, τους καλεσμένους μας, που μας παρουσίασαν τις απόψεις τους και έδωσαν απαντήσεις στον προβληματισμό μας. Πολιτική σημαίνει επιλογές. Πρέπει να κάνουμε πολλές επιλογές οι επόμενες εβδομάδες. Θα κληθούμε να το πραγματοποιήσουμε και εγώ και οι σκιώδεις συγητές. Για παράδειγμα, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη τι είστε κρίσιμο, γιατί ο ίδιος ορισμός του τι είστε κρίσιμο είναι από μόνος του κρίσιμος. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε περαιτέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την εισηγητριά μας. Εν αναμονή της παγκόσμιας διακυβέρνησης ε, και παγκοσμίων κριτηρίων αναφοράς σας επικεντρωθούμε προς το παρόν στα δικά μας, τα ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς, στα ευρωπαϊκά benchmark. Ευχαριστούμε τους καλεσμένους Ράιτ, Σκιάβη, Βαρ, Ζίμπελ και Σάτα. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στη δημόσια κρόση. Τώρα θα διακόψουμε για ένα τέταρτο τη συνεδρίασή μας ε, και θα επανέλθουμε στις 5 ακριβώς για την ε, συζήτηση και ακρόση που θα έχουμε με την Επίτροπο Βέρστεγκερ.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 Merci Paolo. No, Συνάδελφοι, παρακαλώ, καθίστε. για να αρχίσουμε τη συνεδρίαση με το σημείο 8 στην ημερήσια διαταξή. Ανταλλαγή απόψεων με την Μάργαρετ Βέσταγκερ, την επίτροπό μας για θέματα ανταγωνισμού. Να την καλωσορίσω θερμά. Κυρία Βέσταγκερ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που ήρθατε, που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Όπως ξέρετε ήδη, από την ακρόαση κιόλα, η Επίτροπος εξέφρασε την πρόθεσή της να έρχεται εδώ συστηματικά. καθώς και στις συναντήσεις της ομάδας εργασίας για οικονομικές της συνεδρίασής μας για τα θέματα της ανταγωνιστικότητας όπως κατά την ε, πολιτική ανταγωνισμού, την πολιτική κατά τον τραστ, γενικά οτιδήποτε άπτεται της, ε, του ανταγωνισμού. Ε, σας καλωσορίζουμε για αυτή τη θετική σας διάθεση και θα την αξιοποιήσουμε πλήρως. Καλό είναι να μην νομοθεί συνεργασία μεταξύ μας, όχι μόνο γιατί θεωρούμε ότι είμαστε σημαντικό θεσμικό όργανο, αλλά γιατί όντως θέλουμε να ακουστεί και η φωνή των πολιτών τη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων οργανώθηκε για να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό και επίκαιρο θέμα, τη σχέση μεταξύ της συνολικής αξιολόγησης, των τεστ κόπωσε δηλαδή, και των κανόνων ανταγωνισμού, ιδίως για τις κρατικές υπηρετήσεις, και περισσότερο σε ό,τι αφορά τον τομέα, τον κλάδο τον τραπεζικό. Είναι επίκαιρη λοιπόν η συζήτηση, αλλά φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι θα θέσουν και άλλα θέματα. θέματα που ξέρουμε ότι είναι υψηλής προτεραιότητας και ενδιαφέρουν και το κοινό παντού. Φαντάζομαι λοιπόν ότι και η Επίτροπος θα έχει τη διάθεση να συζητήσει και αυτά τα επιπλέον θέματα μαζί μας. Πρώτα απ' όλα θα δώσουμε το λόγο στην ε, Επίτροπο για 10 λεπτά περίπου για την εισηγησή της και μετά θα έχουμε 5 λεπτά για ερωταπαντήσεις με ενδεχόμενες επερωτήσεις αλλά με αρχικό στόχο το 5 λεπτό. Κυρία Επίτροπε, Μάργαρετ έχετε το λόγο. Well, thank you, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν πολύ εγκάρδεο το καλωσόρισμα και περίμενα με ανυπομονησία αυτή την πρώτη μου εμφάνιση στην Επιτροπή σας, την πρώτη ακρόαση μετά την ανάλυση των καθηκόντων. Ελπίζω να είναι η πρώτη από μια σειρά συναντήσεων που θα έχουμε, γιατί άσχετα με τη συνθήκη έχουμε ένα κοινό καθήκον να συνεργαστούμε για να διευρύνουμε τον ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητα υπέρ των πολιτών μας και των επιχειρήσεων. Έχουμε σημαντικές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Δεν χρειάζεται να περιοριστούμε μόνο στα τεστ αντοχής και την αναθεώρηση της ποιότητας του ενεργητικού, ε, την διάσωση με ίδια μέσα ή τις κρατικές ενισχύσεις τράπεζες. Μπορώ να απαντήσω και ερωτήσεις πιο γενικές, αν θέλετε. Δεν χρειάζεται να περιοριστούμε μόνο στον τραπεζικό τομέα. Σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό τομέα και τα αποτελέσματα των δοκιμών αντοχής και την αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικού, θα ήθελα να πω ότι ε, πέρασε ο καιρός της Έχουμε πολλά θετικά αποτελέσματα, αλλά δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμη την κρίση. Δεν έχουμε ακόμη ένα στιβαρό εύρος στο τραπεζικό σύστημα που θα δανείζει σε επιχειρήσεις που έχουν υγιείς επιχειρηματικές ιδέες. Ακόμη πολλοί έχουν παράπονα και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, παραπονιούνται ότι δεν έχουν πρόσβαση σε κεφάλαιο που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν, για να ευημερήσουν. Οπότε έχουμε ακόμη πολύ μακρύ δρόμο μπροστά μας. Τώρα, ποια είναι τα τελευταία στοιχεία από το εργοτάξιο της Τραπεζικής Ένωσης. Στις 26 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τη διεξοδική της αξιολόγηση και με τα τεστ αντοχής ε, δημοσίευσε τα πορίσματα τα αποτελέσματα αυτών των τεστ αντοχής και της διεξοδικής αξιολόγησης. Ε, είχαμε θέματα διαφάνειας και κυρίως του ισοζυγίου των ε, τραπεζών αυτό ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα, μεγαλύτερη διαφάνεια. Και την περασμένη εβδομάδα, στις 4 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέλαβε την ευθύνη να γίνει ε, η ενιαία εποπτική αρχή και να αναλάβει και εποπτικά καθήκοντα στα πλαίσια του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, εποπτικά καθήκοντα επί των τραπεζών. Οπότε έχουμε δύο πολύ θετικέ προοπτικές ε, και πολύ σημαντικά βήματα πρόοδου. Αυτές οι πρωτοβουλίες υλοποιήθηκαν μετά από ετοιμασίες ενός χρόνου και για τον ενιαίο αποπτικό μηχανισμό και για τη δεξαγωγή εκτεταμένων τεστ αντοχής. Εξετάσαμε λοιπόν τους ολογισμούς ε, και την ανθεκτικότητα των μεγαλύτερων τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 130 μεγάλες τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το 80% των συνολικών στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεδομένων των μέτρων ε, ανέβρεση κεφαλαίου που εφαρμόστηκαν από τις τράπεζες ε, μεταξύ ε, Ιανουαρίου και 15 Σεπτεμβρίου μόνο 14 τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν έλλειψη κεφαλαίου, καθαρού κεφαλαίου. 6,5 ε, δισεκατομμύρια ευρώ είναι αυτή, η έλλειψη και αφορά ένα μικρό αριθμό τραπεζών. Πολλές τράπεζες είχαν πρόσβαση σε αγορές ε, την τελευταία χρονιά και φάνηκε γιατί ε, συγκέντρωσαν μεγάλο κεφάλαιο ήταν, ε, παραλαμβάνω, λίγε οι τράπεζε που είχαν έλλειψη κεφαλαίου. Θα πρέπει όμως και αυτό το υπόλοιπο τη έλλειψης κεφαλαίου να καλυφθεί στο ενάμινο που πρόβλεψε η εποπτική αρχή. Και στη φάση αυτή δεν θα πρέπει να προσφύγουν σε κρατικές ενισχύσεις οι τράπεζες ε, όταν έχουν έλλειψη κεφαλαίου αν το ζητήσουν να το κάνουν, κάτι που απευχόμαστε, θα ισχύσουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Πάντως, μέχρι στιγμής η έκβαση ήταν πολύ θετική. Δεν υπευλήθη καμία αίτηση για κρατική ενίσχυση από καμία τράπεζα. Γνωρίζετε, θαυμάσια όπως και εγώ, ότι πριν από ένα χρόνο είχαμε επικαιροποίηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις της τράπεζες ώστε να ληφθούν υπόψη και οι αρχές της Τραπεζικής Ένωσης. Οπότε, αν οποιαδήποτε τράπεζα χρειάζεται να προσφύγει σε χρήματα των φορολογουμένων, οι μέτοχοί της και οι επενδυτές της θα πρέπει πρώτα να συμβάλλουν, ώστε τα κρατικά κονδύλια να είναι πραγματικά το έσχατο μέσο για την, για την ε, συγκέντρωση κεφαλαίου. Σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και τον ανταγωνισμό, εμείς ε, θα μεριμνήσουμε ώστε η χρήση ε, δημοσίων κονδυλίων των χρημάτων φορολογουμένων να παραμείνει στο ελάχιστο απαραίτητο. Θα εφαρμόσουμε τους νέους κανόνες ε, και είναι προφανές ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τα κρατικά κονδύλια και τους φορολογουμένους τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Δεν θα πρέπει να είναι αυτά τα θύματα του ηθικού κινδύνου. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε συνθήκες ίσου ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και να προασπίσουμε και την ακαιρεότητα της ενιαίας αγοράς τράπεζες ε, που θα εξακολουθούν να χρειάζονται δημόσια ενίσχυση θα πρέπει να αναδιαρθρωθούν και να επιστρέψουν ε, στη, στη δανειοληψία από την πραγματική οικονομία. Εκεί θα πρέπει να αναζητήσουν κονδύλια. Θέλουμε μια, ένα υγιές τραπεζικό σύστημα, μπορεί να είναι πιο βαρετό, αλλά ένα τραπεζικό σύστημα που θα επικεντρώνεται στον πρωταρχικό του ρόλο. Ελπίζουμε έτσι να ελαχιστοποιήσουμε τον ηθικό κίνδυνο και νομίζω ότι συμφωνείτε ως προς τη διάγνωση. Χάρη στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και τα σχέδια αναδιάθρωσης και εξυγείας των τραπεζών και χάρη και σε ένα αυστηρότερο και ισχυρότερο, πιο στιβαρό νομοθετικό πλαίσιο και ρυθμιστικό, ο τραπεζικός μας κλάδος έγινε πιο ανθεκτικός και επικεντρώνεται περισσότερο στις ε, βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, δηλαδή στο δανεισμό της πραγματικής οικονομίας ώστε αυτοί που αποταμιεύουν να μπορούν να δανείζουν σε αυτούς που χρειάζονται κεφάλαιο. Φυσικά δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα, έχουμε ακόμη προκλήσει να αντιμετωπίσουμε. Και τα μέχρι τώρα βήματα θα πρέπει ε, να αποτελέσουν το εφαλτήριο για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό τομέα, αλλά δεν θα σταματήσουμε εκεί. Και μετά τα τεστ αντοχής και μετά την ιδιεξοδική αξιολόγηση θα πρέπει να αποδεχτούμε αυτά που κάνουν οι τράπεζες, που θα είναι το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Δεν ε, έχουμε λόγο να είμαστε συγκαταβατικοί να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας. Έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας και οι τράπεζες και το φορολογικό σύστημα. Η αναδιάρθρωση των αδύναμων κρίκων της τραπεζικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη για να μπορέσει να αποκατασταθεί η ρευστότητα κεφαλαίου προς την πραγματική οικονομία. Και φαντάζομαι, συμφωνείτε μαζί μου, ότι ένας υγιής τραπεζικός τομέας αποτελεί το κλειδί για μια υγιή οικονομία. Και αυτό, αυτό χρειαζόμαστε τώρα, ε, έναν ισχυρό τραπεζικό κλάδο που θα πρέπει να διαδραματίζει το ρόλο του στην ε, ευρωπαϊκή οικονομία και να επιστρέψει στο δανεισμό. Φυσικά ε, θα πρέπει προηγουμένως να λάβουμε και κάποια άλλα βήματα. Το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο έχει γίνει πιο στιβαρό από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και φυσικά θα πρέπει τώρα να το εφαρμόσουμε, να λειτουργήσει και αποτελεσματικά, ώστε μετά τη θεωρία να φτάσουμε στην πράξη της Τραπεζικής Ένωσης, να εφαρμοστεί η οδηγία για την αναδιάσταση και την εξηγήση των τραπεζών σε όλα τα κρατημέλη και οι φορολογούμενοι να συνειδητοποιήσουν ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες τους και να μπορέσουν και οι τράπεζες να σταθούν στα δικά τους πόδια, να μην εξαρτώνται από τους κρατικούς λογαριασμούς και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο τραπεζικό τους έργο. Μέχρι στιγμής ήταν πολύ θετικό ότι δεν χρειάστηκαν κρατικές ενισχύσεις στις τράπεζες παρά την έλλειψη κεφαλαίου που είχαν ορισμένε. Και αυτό είναι το βασικό μου μήνυμα. Αυτό το μήνυμα θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σα μεταδώσω σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι μερικοί απουσιάζεται προηγουμένως όταν ο συνάδελφος Τόιρερ ζήτησε από την Επιτροπή ΕΚΟ να συστήσει μια προσωρινή εξεταστική επιτροπή για να διερευνήσει θέματα φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και φορολογικής απάτης επευκαιρία των πρόσφατων διαρών για το σκάνδαλο στο Λουξεμβούργο. Εγώ ολόθερμα και ολόψυχα είμαι υπέρ τη ε, σύσταση μια τέτοια επιτροπή. Και θα ζητούσα και από την αρμόδια επίτροπο ανταγωνισμού να προχωρήσει περαιτέρω τι έρευνε για το θέμα αυτό. Και σε σχέση με την αυριανή συζήτηση, μα εξέπληξε το γεγονό ότι έπαψε να έχει το χαρακτήρα κρατικών ενισχύσεων. Ε, και θα ήθελα να το σχολιάσετε ευκαιρία για τις παρουσίες του κ. Μοσκοβισή. Θα ήθελα πάντως να σας καλωσορίσω στην πρώτη σας αυτή εμφάνιση στην ε, Επιτροπή ΕΚΟΝ, κυρία Φεστάγκερ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού ε, με βάση τον νέο μηχανισμό, ε, νέο, μηχανισμό Θα πρέπει οι αποφάσεις να λαμβάνονται σε πολύ στενόχρονο διάγραμμα και οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να είναι νομικώς ανεπίληπτες. Πιστεύετε ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού θα ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της σε τόσο πιεστικά χρονοδιαγράμματα. Τι ειδικά μέτρα θεσπίσατε και πώς λειτουργούν οι εσωτερικές διαδικασίες της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης ώστε οι αποφάσεις που θα κληθεί να, λάβει με, βάση τον ενιαίο μηχανισμό εξυγείας θα, είναι, θα λαμβάνονται σύντομα και θα είναι αντικειμενικές και νομικώς ε, άψογες. Ευχαριστώ. Τώρα μόλις ενημερώθηκα για την πρότασή σας να συστηθεί ειδική εξεταστική επιτροπή με θέμα την φοροδιαφυγή, φόρο και φορολογική απάτη. Και θα πρέπει να διαμορφώσουμε μια πλήρη εικόνα, γιατί εγώ το βλέπω αυτό υπό το πρίσμα του ανταγωνισμού. Αλλά υπάρχει και ένα γενικότερο ζήτημα φορολογικής νομοθεσίας και γι' αυτό προηγουμένως ανέφερα την πρόταση της κοινή ενοποιημένης φορολογικής εταιρικής βάσης. Ένα θέμα που θα μπορούσε να απασχολήσει ενδεχομένως μια τέτοια ειδική επιτροπή. Και σίγουρα και τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να συμβάλλουν στο έργο αυτό. Γιατί υπάρχει μια λεπίδραση μεταξύ της εθνικής φορολογικής νομοθεσίας, των δικών μας προσπαθειών για τις κρατικές ενισχύσεις και ε, τον ανταγωνισμό και τη λειτουργία των ε, διατάξεων αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τα φορολογικά θέματα απαιτείται ομοφωνία στο Συμβούλιο και θα δούμε ποια θα είναι η ταχύτητα της πρόοδου. Δεν νομίζω ότι εγώ είμαι πιο αισιόδοξη από, από σας. Βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν θα αποφασίσουμε, εγώ δεν δεν είναι δική μου αρμοδιότητα πώς θα οργανώσετε την εντολή αυτή της Ειδική Επιτροπή, αλλά φαντάζομαι μπορούν να συμβάλλουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και συμφωνώ ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και εγώ θα έχουμε λόγο στο μέλλον και για το θέμα του ενιαίου μηχανισμού. Το ίδιο θα κάνουν και οι εποπτικές αρχές με βάση τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό θα εξετάσουν θέματα κρατικών ενισχύσεων, ε, η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα επίσης, για να επικεντρωθούμε μόνο σε ένα σημαντικό ζήτημα. Εμείς θα φροντίσουμε να έχουμε τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητες να αναλάβουμε το έργο μας. Και συμφωνώ ότι η ταχύτητα ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ. Πάντως, ακόμη και όταν ήταν πιο επιτακτική η ανάγκη και πιο επίγουσα η κατάσταση όταν σοβούσε η κρίση δεν υπήρχε πρόβλημα. Το θέμα είναι να εξασφαλίσουμε και πόρους αλλά και τις απαραίτητες γνώσεις για να δράσουμε με ταχύτητα. Πάντως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Από την... Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε για την ε, θαυμάσια προφορά του ονόματός μου. Όχι, πραγματικά το εννοώ το κομπλιμέντο. Να ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Luxembourg Λίξ, Juncker ε, Λίξ. Επίτροπε, είπατε ότι πολλά από τα στοιχεία για... που γίνονται στο Λουξεμβούργο ενδεχομένως να είναι νόμιμα. Αυτό αποτελεί την ουσία του προβλήματος. Είναι κοινικό και εξοργιστικό. για ένα τρισεκατομμύριο που χάνεται από φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και τίθονται θέματα δαπανών κρατικών, υποδομές κτλ. Είπατε ότι ενοποιήσατε την ε, εταιρική φορολογική βάση χωρίς μια ελάχιστη φορολόγηση που δεν επιτρέπεται με τις συνθήκες αυτό μπορεί ακόμα να κάνει πιο έντονη την, τον ανταγωνισμό μεταξύ φορολογικών συστημάτων. Ερωτήσεις λοιπόν έχω να σας κάνω. Η συμμόρφωση του Λουξεμβούργου, η συνεργασία με την ε, Επιτροπή είναι καλύτερη από τότε που δεν είναι στη θέση του. Δεν έχει αξίωμα ο κύριος Γιούγκερ. Σύμφωνα με τους, τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με συλλογική ευθύνη. Πώς θα διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του κυρίου Γιούγκερ. Πώς θα τα καταφέρετε. Και τρίτη ερώτηση αν υπάρξει αγωγή κατά του Λεξεμβούργου και μπορέσετε να αποδείξετε ότι υπήρξε προνομιακή μεταχείριση των επιχειρήσεων αυτών και ξεκινήσει η έρευνα. Πιστεύετε ότι ο κύριος Γιούγκερ θα εξακολουθήσει να είναι κατάλληλος για τη θέση αυτή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας ζητώ να απαντήσετε με ένα ναι και με ένα όχι. Ή να σας το πω αλλιώς, ότι αν έπρεπε να το αφιερώσετε ένα τραγούδι, ποιο θα το αφιερώνετε, το Ζωνερή αντί της Edith Piaf, το I Did My Way ή ποιο άλλο τραγούδι. Κύριε Επίτροπε, θα σας ε, παρακαλέσω να μην με προκαλέσετε να τραγουδήσω θα έρθετε σε δύσκολη θέση. Καταρχάς, είναι διαφορετική η αξιολόγηση της κοινή ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις επιχειρήσεις. Εγώ πιστεύω ότι θα βοηθούσε. Και εγώ θεωρώ ότι θα βοηθούσε τις επιχειρήσεις που δεν κάνουν φορολογικό προγραμματισμό να πληρώνουν το φόρο που πρέπει να πληρώνουν χωρίς να χρειάζεται να απασχολούν διάφορους φορολογικούς δικηγόρους σε διάφορες χώρες προκειμένου να το κάνουν αυτό με σωστό τρόπο. Αυτό ασφαλώς ε, είναι υποκειμενικό στοιχείο και υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Ναι, ε, είδαμε καλύτερη συνεργασία με το Λουξεμβούργο. Εγώ δεν ε, εικάζω το γιατί, τα αίτια. Αλλά πολύ χαίρομαι που απλά συνέβη αυτό, γιατί πολύ απλά διευκολύνει το έργο μας. Αυτό για την πρώτη σας ερώτηση. Κατά δεύτερον, για τις νέες έρευνες. Ως τώρα είχαμε πάρει την απόφαση να, να ανοίξουμε τέσσερις ε, έρευνες μετά από μία προκαταρτική έρευνα. Οι πιο πολλές εξ αυτών, οι δύο από τις τέσσερις αποφάσεις, είναι δημόσιες πλέον. Η τρίτη θα δημοσιευθεί σε λίγες ημέρες προκειμένου να δούμε ποιες ήταν οι προκαταρτικέ έρευνες και γιατί δικαιολογούν την ε, έναρξη επίσημης έρευνας. Εγώ δεν άκουσα ούτε έχω ακούσει, ούτε έχω δει κάτι που θα μου έδινε τα χέρια. Αντιθέτως, αυτό που έχω δει και έχω ακούσει και αυτή είναι η εντύπωση που θέλω να σας δώσω ότι έχω το ελεύθερο να κάνω ό,τι πιστεύω καλύτερο στην προκειμένη περίπτωση. Κατά τρίτον, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην νικάζω. Για κάποιες επιχειρήσεις είναι πολύ άβολο να διαπιστώσουν τι φόρους θα πληρώσουν σύμφωνα με τις αποφάσεις. Το πρόβλημα είναι αν οι αποφάσεις προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού, αν επισέλθουν στον τομέα της κρατικής ενίσχυσης. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Και γι' αυτό δεν ε, δαπάνω το χρόνο μου κοιτώντας ε, προσωπικότητες ε, και θεωρώ ότι στη δημόσια συζήτηση πρέπει να συζητάμε τους φόρους και τα φορολογικά ζητήματα, τη στρέβλωση του φόρων και όχι προσωπικά ζητήματα. Ευχαριστώ κύριε Δράιμερ από τους Πράσινους τώρα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Επίτροπο. Είμαι ο έκτος της σειρά ομιλητής και υποφελούμε από το πλεονέκτημα, δεν χρειάζεται να επαναλάβω. μας λέτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μας λέτε για τα σχέδιά σας για την επόμενη πενταετία. Αυτό σας ρωτώ λοιπόν. Είπατε θα λάβετε υπόψη τις νέες πληροφορίες που διέρευσαν από το Wikileaks. Δεν αρκεί αυτό. Προτίθεστε μέσα στην πενταετία της θητείας σας να πραγματοποιήσετε και έρευνες ώστε κατά το πέρας της θητείας σας πιστεύετε ότι το ευρωπαϊκό φορολογικό σύστημα ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα της φοροδιαφυγής, να ελέγχεται η φοροδιαφυγή από, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊκό επίπεδο πλήρως ε, και ολοκληρωτικά. Είναι αυτός πολιτικός σας στόχος. Είπατε ότι είστε υπέρ μιας ε, ενοποιημένης φορολογικής βάσης. Είστε υπέρ ε, της ενημέρωσης αναχώρα, ε, φορολογικής ενημέρωσης αναχώρα για τις πολυεθνικές εταιρείες. Είναι και αυτός ένας πολιτικός σας στόχος. Ε, ήσταν αρκετά αόριστοι στην, στο σχολιασμό της πολιτικής του κυρίου Γιούγκερ. Θεωρείτε ότι τέτοιου είδους φορολογικά ε, σχέδια και συμφωνίες φοροαποφυγής ε, μεταξύ πολυεθνικών και κυβερνήσεων δεν θα πρέπει να έχουν τη θέση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη πενταετία. Ευχαριστώ. Η Επιτρόπος έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Οι ερωτήσεις σας ε, προδίδουν μεγάλη εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου. Θα πρέπει όμως να είμαι κάπως πιο σεμνή και ταπεινή, γιατί έχοντας παρακολουθήσει τις προηγούμενες προτάσεις ε, του Επιτρόπου ΣΕΜΕΤΑ για τα φορολογικά θέματα και έχοντας παρακολουθήσει και τη συζητήση στο Συμβούλιο για θέματα φορολογικής πολιτικής, αποκόμισα την εντύπωση ότι είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε αμοφωνία στο Συμβούλιο για να σημειώσουμε πρόοδο σε φορολογικά ζητήματα. Και ακόμη κι αν συσπυρώσουμε τις προσπάθειές μας και συνταχθούμε Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες για να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι χρειαζόμαστε κάποιες κοινέ διατάξεις για την φορολογία των εταιριών στην Ευρώπη. Δεν θέλω να αποφύγω τη συζήτηση. Σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν θα πρέπει η συζήτηση αυτή να μονοπολίσει το θέμα αυτό να πονοπολίσει τη συζήτηση και να αποσπάσει την προσοχή μας από άλλα θέματα που είναι σημαντικά, όπως είναι η ολοκλήρωση των εκκρεμών υποθέσεων, η διαμόρφωση πιο τεκμηριωμένης γνώμης για το τι συμβαίνει και με τις γνώσεις αυτές θα λάβουμε αποφάσεις για το τι μελγενέστε. Και δεν αποφεύγω τη συζήτηση, αλλά θέλω να βρούμε έναν αποτελεσματικό τρόπο για να καταλήξουμε σε αποτελέσματα και να μην έχουμε διάξει των προσπαθειών μας, αλλά να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα θέματα με διαρθρωμένο τρόπο και να διεκπαιρώσουμε τις εκκρεμότητες, τις εκκρεμείς υποθέσεις και μετά από αυτό να αποφασίσουμε αν θα ξεκινήσουμε και νέες, που κατά πάσα πιθανότητα θα το κάνουμε. Τους μη ο Αργανόπουλος. Κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για τα στρέστες τεστ των τραπεζών. Την, κατάσταση, την κακή κατάσταση του ελληνικού λαού τη γνωρίζετε και γνωρίζετε βέβαια ότι τώρα η Τρόικα, δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση ρυθμίζουν τα καθυστερούμενα τραπεζικά δάνεια. Με μοναδικό κριτήριο το κέρδος των τραπεζών και κατά τη δικιά τους κρίση και μόνον ρυθμίζονται μόνο τα δάνεια των βιώσιμων όπως λέγονται επιχειρήσεων, δηλαδή των μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν και οι αυτοπασχολούμενοι εξαιρούνται και οδηγούνται σε κλείσιμο. Από τα στεγαστικά δάνεια ανέργων μισθωτών δεν κουρεύεται ούτε ένα ευρώ. Το πολύ πολύ δίνεται μία παράταση εξόφλησης κοροϊδία διότι ε, όπως γνωρίζετε και η ανεργία και η μισθή θα διαρκέσουν, η χαμηλή μισθή πείνα θα διαρκέσουν για πολλά χρόνια από μία πρώτου του 2015 ξαναρχίζουν οι πληστηριασμοί σπιτιών και χιλιάδες κόσμος θα χάσει τα σπίτια του. Ξέρετε, όλα αυτά είναι προϋποθέσεις για να περάσουν τα, τα stress test τράπεζες στην Ελλάδα και παντού. Τελικά, τη θέση των μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων θα τις λάβουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, γη και ακίνητα θα περάσουν σε μεγάλα συμφέροντα. Ε, εμείς λέμε ότι τελικά αυτή η ανταγωνιστικότητα οφείλει μόνο τους μεγάλους. Εσείς τι λέτε, και ιδιαίτερα τι λέτε για την έναρξη των πληστηριασμών στην Ελλάδα από 1 πρώτου 2015 όπου χιλιάδες κόσμος θα χάσει τα σπίτια του. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ίσως να βλέπω λίγο διαφορετικά τα γεγονότα και τα στοιχεία που προέκυψαν από τα τεστ, από τα τεστ κόπωσης για την αξιολόγηση των στοιχείων ενεργητικού. Εγώ βλέπω ότι ο τραπεζικό κλάδο είναι υγιέστερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο, διότι συγκεντρώθηκε αρκετό κεφάλαιο και μόνο ένα μικρό αριθμό τραπεζών, σε 8 κράτη-μέλη 13 τράπεζε, είχαν έλλειμμα στο κεφαλαίο του. Καμία δεν ήρθε να μα πει θέλουμε κρατική βοήθεια. Αυτό είναι ήδη θετική εξέλιξη. Δεν αλλάζει την κατάσταση βεβαίως για τις ε, οικογένειες, τις επιμέρους στην Ελλάδα. Αλλά το να έχουμε βροστότερο γέστρο τραπεζικό σύστημα ίσως να ωφελήσει αυτό έπειτα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι ο τραπεζικός και ο χρηματοπιστωτικός κλάδος θα διαμαντήσουν το λόγο τους για την οικονομία και θα μπορέσουν οι άνθρωποι να ε, χρηματοδοτήσουν τις νεοφύης επιχειρήσεις τους, να συγκεντρώσουν κεφάλαιο για να κάνουν κάτι. Αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι θα δούμε φως στην άκρη του τούνελ. Ακόμα και αν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ιδίως νέοι, που το βλέπουν αυτό πολύ μακρινό. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με το Ευρωπαϊκό Λογικό Κόμμα, η Έστρε Ντελάνγκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. σα ευχαριστώ, Επιτροπέ, που βρίσκεστε εδώ και που θέλετε να επιτύχετε ανοιχτό πνεύμα για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Είσαστε πάρα πολύ συνοπτικοί. Κάνετε κάποιε διακρίσει και επιμένετε για να εξαντλήσετε τα θέματα αυτά, που είναι πολύ δύσκολα, αλλά πολύ επανερχόμαστε στο θέμα τη φοροαποφυγή φοροδιαφυγής. Γιατί βλέπουμε την αδικία και την αγανάκτηση των Ευρωπαίων πολιτών όταν βλέπουμε αυξημένο φορτίο φορολογίες και βλέποντας ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα να περάσουν τα σύνορα και να φτιάξουν, να μαγειρέψουν ε, ένα σύστημα αντί να πληρώσουν τους φόρους που όλοι πληρώνουμε. Αυτή η αδικία, αυτό το αίσθημα αδικίας λοιπόν είναι που ε, μας απασχολεί. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν που αισθάνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες και που εκφράζουν στη συζήτηση αυτή. Θα ήθελα λοιπόν, γιατί είπατε ότι οι πληροφορίες πλάνα είναι δημόσιες, χάρη στους δημοσιογράφους και ότι αυτές δεν είναι όλες οι πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε πιο πολλά από τις εθνικές αρχές. Ξέρω ότι στη δική μου χώρα, στην Ολλανδία, είναι μέσα σε αυτές τις δομές αυτές και οι αρχές, οι φορολογικές υπηρεσίες δεν σας δίνουν τις πληροφορίες αυτές, δεν το δίνουν ούτε καν στο Εθνικό Κοινοβούλιο τις πληροφορίες αυτές. Συμφωνώ λοιπόν ότι οι τέσσερις αυτές υποθέσεις θα σας βοηθήσουν να αναλύσετε αυτά που γίνονται στην παρούσα φάση, αλλά η γνώση θα έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο Και θα δημιουργηθούν νέε ε, δομές. Θα χρειαστεί λοιπόν να τρέχουμε πίσω από την πραγματικότητα πάντα, γιατί συνέχεια θα δημιουργούνται, θα, θα βρίσκονται νέα συστήματα. Τι θα κάνουμε λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι εδώ μέσα που λένε ότι οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να δημοσιευθούν από την αρχή μέχρι το τέλος, από το α μέχρι το ω, κάθε τελεία, κάθε κόμμα. Δεν συμφωνώ απαραίτητα. Πιστεύω ότι υπό τους ε, κατάλληλους όρους ε, τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να γνωρίζουν την ουσία των ε, αποφάσεων για να καταλάβουν τι συμβαίνει. Και συμφωνώ ότι αν δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, δεν μπορούμε να προτείνουμε οποιαδήποτε λύση στο πρόβλημα. Αυτό λοιπόν θα σας ήταν ωφέλιμο στο εσωτερικό των εθνικών αυτών ε, αποφάσεων. Η κυρία Επίτροπος έχει το λόγο. Ναι. Μία εκ των έσω διάσταση της ευρωλογικής απόφασης θα μας δώσει μία αίσθηση δομικής, διαστατικής προσέγγισης. Καταλαβαίνω ασφαλώς γιατί αυτό συζητιέται και γιατί υπάρχουν και διαφωνίες. Προφανώς οτιδήποτε δημοσιεύεται, αποτελεί αντικείμενο συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι είναι ίσως και υπερβολικό να πούμε ότι κάθε δικαστική απόφαση θα πρέπει να δημοσιευτεί. Ναι, ναι, ναι, δεν το είπατε αυτό και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, γιατί υπάρχει το θέμα του απορρίτου. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία που πρέπει να προστατεύσουμε, προκειμένου να μπορεί ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Αλλά για μας θα είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε, να γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις ε, για τα φορολογικά ζητήματα. Ένας από τους λόγους που με κάνουν να πιστεύω ότι θα μπορούσαν να ήταν ε, χρήσιμοι εταίροι τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι ακριβώς αυτός. Γιατί στην περίπτωση αυτή θα αποτελούσε ένα τόπο όπου θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν ισορροπημένο διάλογο να κάνουμε μια καλύτερη δημόσια συζήτηση για τους φόρους, τα προλογικά συστήματα, τη φοροδιαφυγή και τον προλογικό ανταγωνισμό που βλέπουμε στην Ευρώπη. Γιατί ακόμα και επισήμω ο εταιρικό συντελεστή φορολόγηση είναι πολύ διαφορετικό από κράτο μέλο σε κράτο μέλο. Άρα ναι, αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα σύστηνα ένθερμα. Ευχαριστώ από του σοσιαλδημοκρατέ τώρα. Ο κύριος ε, Τζάνι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, να σας εκμυστηρευτώ. Είμαι καινούριο βουλευτής. Ίσως να μην είμαι τόσο γνώστης όσο κάποιοι συνάδελφοι εδώ. Αλλά δεν είμαι και αφελής ταυτόχρονα. Οπότε, ήθελα να γύρω κάποια από τα ζητήματα που και σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται αντιληπτά α, ε, ως αρκετά σημαντικά. Το ίδιο και στη χώρα μου την Ουγγαρία. Το σκεφτόμουν, το σκεφτόμουν πολύ αυτό για το Λουξεμβούργο, το Luxembourg Leaks. Και δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες και στα πράγματα που έγιναν το παρελθόν, αλλά εγώ ως ταπεινός Ούγγρος, έστω και βουλευτής, κάτι που είναι πολύ πιο ευχάριστο βέβαια, θα προτιμούσα να ε, πληρώνω φόρο στο Λουξεμβούργο από ότι οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Είναι προφανές. Και αυτό το λέγαμε κάποτε ως μύθο. Τώρα τι βλέπουμε, ισχύει. Οπότε για την ερχόμενη πενταετία, ή τέλος πάντων 4,5, τα 4,5 χρόνια που έρχονται, το να μην βρεθούν νομικοί πολιτικές αποκρίσεις για το παρελθόν είναι κάτι, αλλά για το μέλλον κάτι πρέπει να κάνουμε. Έχω στείλει μια-δυο επιστολές στην προηγούμενη επιτροπή και η απάντηση ήταν πάντοτε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ο κανόνας. Μα η ερώτησή μου είναι η εξή. Εάν η αντίληψη του κοινού βασίζεται σε, αποφασίζει για κάτι ότι δεν είναι καλό, ε, δεν πρέπει κάτι να αλλάξουμε. Έστω και στους κανόνες. Καταλαβαίνω. Και το αντιλήφθηκα με τις ε, πολλαπλές ακροάσεις των διαφορών επιτρόπων. Ότι η φορολογία θα μπορούσε να είναι κάτι ότι η φορολογία είναι κάτι που δεν μπορεί να αγγίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι τελείω στα πλαίσια των νομοθετήτων των κυβερνήσεων. Αυτό το μήνυμα ήταν σαφέ, παρά τι ε, περίπλοκε κάποιε φορέ απαντήσει και διαλόγου. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και ίσω και το Συμβούλιο, είναι να εντοπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα. Ένα από τα δικά μου τα προβλήματα είναι ότι η φορολογία είναι τόσο διαφοροποιημένη ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα παράδειγμα για τα τρόφιμα. Σε κάποιες χώρες είναι μηδενική η αξία κάποιων προϊόντων. Στη δική μας να ε, μας 27 ε, ευρώ. Δεν είμαστε ίσοι με τους υπόλοιπους. Λοιπόν, είναι πολλά αυτά που θα πρέπει να συζητηθούν, αλλά πρώτα απ' όλα Εάν μπορείτε να επηρεάσετε και να περιορίσετε τη διαφθορά, έχοντας κατά ότι η διαφθορά δεν είναι μόνο εταιρική, αλλά κυβερνητική, θα ήταν κάτι. Μια πολύ σύντομη παρατήρηση από μένα τον ίδιο, αν επιτρέπετε. Εάν θέλετε απάντηση από την Επιτροπή, θα ήταν καλό να κάνετε και συγκεκριμένη ερώτηση. Είναι και πιο εύκολο για την ίδια μετά. Κοιτάξτε, για κάθε νεοβουλευτή έχω μεγάλο σεβασμό γιατί και εγώ ίδια νέα επίτροπος είμαι. Απλώς να πω το εξή γιατί κάποιε φορέ νομίζω ότι οι ένομες ε, αντιδράσει για το παρελθόν ίσως να ήταν και γέφυρα για να βρούμε τις πολιτικές αποκρίσει για το μέλλον. Γιατί έτσι γίνεται κάνει συνετότερος. Έτσι καταλαβαίνει πώ λειτουργούν τα πράγματα. Και βάσει αυτής της υπόθεσης μπορεί κανείς τελικά να αλλάξει και το πώς συζητούνται τα θέματα δημοσίως και την προσέγγιση όλων σε αυτά. Εδώ χρειάζεται μια πολύ στενή συνεργασία, μια πολύ στενή ε, μια κοινή προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Από την πλευρά τη Επιτροπή μπορούμε να κάνουμε αυτό που είναι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μα, τίποτε παραπάνω. Αλλά ε, τα φορολογικά ζητήματα είναι σοβαρότατα από ό,τι φαίνεται. Οπότε πρέπει να συζητηθούν και στο Συμβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Σε αυτές τις συνθήκες μόνο θα προχωρήσει ο δημόσιος διάλογος και θα πετύχουμε αλλαγές. Θυμηθείτε απλώς ότι μπορέσαμε να έχουμε την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τα εισοδήματα που έχουν ε, κερδιθεί σε άλλη χώρα από όπου φορολογείται κανείς, κάτι που δεν θα μπορούσαμε καν να το διανοηθούμε θα το είχαμε πετύχει πριν από πέντε χρόνια. Τώρα το κάναμε. Η αλλαγή γίνεται μόνο αν υπάρξει αυτή η στενή συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Μάτος Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ελπίζω Η, τα στιγμιότυπα αυτά που είδατε και τα όπως να ήταν ευχάριστα. Εγώ θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Στην γενική σας διεύθυνση είδατε τις προάλλες εργάτες από τη Χαλιβουργία της Τέρνη. Ε, και είναι θεαματικό πως η Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία τελικώς καταστρέφει συχνά την οικονομία αντί να ευνοεί την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ας θυμηθούμε ότι αυτή η Χαλιβουργία πωλήθηκε στους Φινλανδούς του Οτοκούμπου και μετά από την αγοραπολισία αυτή έκλεισε. Διότι έχουν δεσπόζουσα θέση οι Φινλανδοί και τελικά επέστρεψε στην Τίσεν, στον όμιλο Τίσεν, η ε, Χαλιβουργία. Και τελικά έτσι ανακοινώθηκαν 153 απολύσεις γιατί έχει ένα κοινωνικό πρόγραμμα ο Όμιλος Τάισεν. Τώρα έχουμε τόσες ασιατικές ε, χαλιβουργίες, τόσες ασιατικές εταιρείες. Και μιλάμε για δεσπόζουσα θέση, για κανονισμούς και διατάξεις που ανήκουν στο παρελθόν. Πριν από μία εβδομάδα ε, έγιναν δεκτοί οι εργάτε στη γενική σα διεύθυνση. Εγώ σα ρωτώ αν υπάρχουν εξελίξει, αν έχετε κάποια είδηση για το σημείο αυτό. Διότι 153 Ιταλικέ οικογένειε περιμένουν μια απάντηση. Περιμένουν μια απάντηση από μια Ευρώπη που όταν συμπεριφέρεται έτσι του φαίνεται πραγματικά πολύ απομακρυσμένη και πάρα πολύ αδιάφορη προ το δικό του πρόβλημα. Η Επίτροπος παρακαλώ. Ελπίζω να συνειδητοποιήσετε ότι έχουμε ως κοινό στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Μερικές φορές βέβαια δεινοπαθούν οι επιχειρήσεις και χάνουμε θέσεις απασχόλησης και χρειάζεται χρόνος για να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης σε άλλους τομείς ή να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις. Για το συγκεκριμένο θέμα ελήφθησαν αποφάσεις και τα μέτρα που προτάθηκαν για την συγχώνευση αυτή των επιχειρήσεων έγιναν δεκτά. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι την οδύνη που προκάλεσε αυτή η απόφαση και προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Ελπίζω να το κάνουμε από κοινού με τους ε, ιδιοκτήτες ε, της επιχείρησης. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, κάναμε ό,τι μπορούσαμε με βάση τους κανόνες του ανταγωνισμού πέρασε το θέμα από εμά και ξεκινά η φάση για τις επιχειρήσεις. Θα γίνει αναδιάρθρωση και αυτό θα το αναλάβει η επιχείρηση. Ευχαριστώ. Η Ανελίζε Ντότς για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Και εγώ νέα Ευρωβουλευτής είμαι και θα ήθελα να σας ξανακαλωσορίσω θερμά στην ε, Επιτροπή μας μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας και προσβλέπω σε συνεργασία για να βρει φάσμα θεμάτων. Θα επανέλθω όμως στο βασικό θέμα, τη σχέση φορολογίας και ανταγωνισμού. Άκουσα με προσοχή όλες σας τις απαντήσεις. Κατά τη γνώμη μου, τρία θέματα μένουν εκκρεμή. Χρειάστηκαν 80 δημοσιογράφοι και ένα εξάμεινο για να αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες και να δημιουργηθεί αυτή η διαρροή για το σκάνδαλο του φοροαποφυγής στο Λουξεμβούργο. Και φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακαλύπτει λεπτομέρειες από τον τύπο, από τις εφημερίδες, αντί να τις συγκεντρώνει με δικές της έρευνες. Πώς με έμπρακτο τρόπο θα συνεργαστείτε με τον Επίτροπο Μοσκοβιτσί και τις αρμόδιες διευθύνσεις σας για να πατάξετε αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή Επίσης, ε, πώς θα, εγκρι... ενθαρρύνετε την, ε, ε, γενική σας διεύθυνση για να αναλάβει μέτρα και να δράσει δημιουργικά και με πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσει τέτοια θέματα φοροδιαφυγής και να διερευνήσετε τις υποθέσεις. Πολλά μας είπατε για την προβληματική σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και και κρατών και την συγκαλυμμένη μορφή κρατικών επενδύσεων. Μερικές ε, ε επιχειρήσεις εφόσον καταβάλουν σχεδόν μηδενικούς φόρους δεν θεωρείται ότι, είναι εγενός, ε, δεν θεωρείται ότι εγενός στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Έχουμε μεγάλη οικονομική κρίση και μικρές εταιρείε τριμώχνονται και χρεοκοπούν γιατί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις μεγάλες πολυεθνικές ε, που εποφελούνται από φορολογικές απαλλαγές και οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ε, φορολογικά τις μεγάλες πολυεθνικές που στην ουσία δεν καταβάλουν καθόλου φόρο. Θα ήθελα λοιπόν να σας απευθύνω παράκληση θερμή να πρωτοστατήσετε σε θέματα ανταγωνισμού και να στρέψετε τη συζήτηση και σε φορολογικά θέματα. Γιατί δεν είναι θέμα που αφορά μόνο τι κρατικέ ενισχύσει αυτή η φορολογία, αλλά και τον ανταγωνισμό. Αφορά άμεσα τον ανταγωνισμό, γιατί τέτοιε φορολογικέ πρακτικέ ε, θίγουν και πλήττουν ανεπανόρθωτα τον ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία για να σημειωθεί πρόοδο είναι η συνεργασία με τα κρατη και να λάβουμε τις πληροφορίε που ζητάμε από τα κράτη-μέλη. είναι και ο λόγος όπως αναφέραμε και προηγουμένως, που έχουμε ζητήσει από κάποια κρατημέλη να μας παρέχουν πολλές πληροφορίες. Κάποιες ε, χώρες έχουν επιδείξει κάποια προθυμία, πώς να το πω. Τόσο απρόθυμες φάνηκαν που ζητήσαμε από το δικαστήριο να τις αναγκάσει να μας δώσει τα στοιχεία που ζητάμε. Ευτυχώ έχει βελτιωθεί έκτοτε η συνεργασία και ελπίζω ότι θα βελτιωθεί περαιτέρω. Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον όλων να είναι στενή η συνεργασία με τα Αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο. Γιατί μεταλαμβάνουμε τις πληροφορίες, λαμβάνουμε κάποιες πληροφορίες από την δημοσίευση των σχετικών εγγράφων και αυτό που θα πρέπει να κάνω είναι να συνεχίσω αυτή την task force για τα φορολογικά αυτή την ομάδα δράσης, η TAX Task Force, να συνεχίσει τη συνεργασία με την DG ε, Comp για να μην είναι μόνη της η ομάδα δράσης αυτής και να συλλέξει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Προκειμένου να τους προσθέσουμε πόρους όπου χρειάζονται. Είναι κάπως ενοχλητικό, το ξέρω, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνουν διαθωμένα βήματα για να είμαστε πιο ευφυείς, να συλλέξουμε εμπειρίες. Τι κάνουμε με τις τέσσερις ανοιχτές ε, υποθέσεις, για τις δύο εξ αυτών έχουν δημοσιευθεί στοιχεία, για την τρίτη θα δημοσιευθούν συντόμως, μέσα στην εβδομάδα και έτσι, τρίτη θα μπορέσουν να σχολιάσουν την ανοιχτή αυτή έρευνα. Και έτσι θα μπορέσουν να διεξαχθούν οι έρευνες πιο γρήγορα. Καταλαβαίνω λοιπόν τι λέτε και συμφωνώ με την εκτίμησή σας. Αλλά έχουμε αποδεχτεί ότι υπάρχει νόμιμη τέτοια τέτοιος ανταγωνισμός για τα φορολογικά ζητήματα και έχουμε αποδεχτεί ότι χρειάζεται και μοφωνία για να αλλάξει αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι έχουμε ακόμα πολλή συζήτηση μπροστά μας. Ευχαριστώ. Ο Βέρνερ για το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω κυρία Επίτροπε για τον διορισμό σας. Έχουμε όχι μόνο μεγάλη εμπιστοσύνη, αλλά έχουμε να αποθέσει και μεγάλες προσδοκίες πάνω σας σε ό,τι αφορά την ενεργό προάσπιση της φορολογική πολιτικής. Γιατί η φορολογική πολιτική δεν είναι τόσο αγαπητή όσο θα έπρεπε σε μια οικονομία τέτοια, στην κοινωνική οικονομία. Γι' αυτό λοιπόν επαφιόμαστε στην ε, δράση σας. Έχω μεγάλη εμπειρία και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να επανέλθω σε δύο υποθέσεις, σε δύο αποφάσεις που έχουν ληφθεί καταρχάς η διστακτική στάση του Επιτρόπου σε ό,τι αφορά το θέμα της Google. Όλοι ξέραμε ότι ότι χρειάζεται απόφαση καταπηγόντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση της ε, θέσης εξουσίας. Ο κ. Αλμούνια ήταν απρόθυμος. Δεν θέλουμε να δακτυλοδείξουμε οποιοδήποτε, αλλά θέλουμε να κοιτάξουμε το μέλλον. Και ύστερα τι θα γίνει στο μέλλον της ε, νομικής διαμόρφωσης του συστήματος του προλογικού, Το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο διαδικασίας ε, συναπόφασης μπορεί να συμπεριληφθεί προκειμένου να κρίνουμε για τους κανόνες de και για άλλες πολιτικές βασικές αρχές που νομιμοποιούν τη δική σας πολιτική. Θα νομιμοποιούσαν πολύ τη δική σας πολιτική. Και μεταξύ και σε αυτά συγκαταλέγεται και αυτό που δεν ε, αποφασίστηκαν. Εντυπωσιακές περιπτώσεις ε, κρατικών ενισχύσεων, πάνω από 500 εκατομμύρια για την Eurocrane για παράδειγμα, στι 30 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν τη λήξη της θητείας του, μία μέρα πριν τη λήξη της θητείας του, μου έγραψε τις αποφάσεις, τα επιχειρήματα που υποστήριξαν την απόφαση που είχε λάβει πρώτη Οκτωβρίου. Θα ήθελα να εξετάσετε τα επιχειρήματα αυτά και ενδεχομένως να τα αναιρέσετε. Γιατί όλα έγιναν υπερβολικά εσπευσμένα τελευταία στιγμή. Και δεν νομίζω ότι ήταν θετική η απόφαση. Σας ευχαριστώ. Η Επιτρόπος έχει το λόγο. Νομίζω τέθηκαν τρεις διαφορετικές ερωτήσεις. Και όχι δύο όπως αναγγέλθηκε. Ελήφθη απόφαση. Και για να είμαι ε, σαφής, δεν ε, μπορώ να σα την... Ε, δεν μπορώ να πω περισσότερα τώρα. Ε, όσο για το Κοινοβούλιο θα πρέπει να βρίσκεται πιο μπροστά από την νομοθεσία. Για τις κρατικές επιδοτήσεις λόγω χάρη έχουμε ήδη εξελαχίστων ε, κανόνες και εξαιρέσεις συνολικές, αλλά θα προκύψουν και άλλα θέματα με τη Λευκή Βίβλο και ούτω καθεξής. Οπότε θέλω να είμαστε συγκεντρωμένοι και να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση για τα θέματα αυτά πριν πάρουμε το χαρτί και το στυλό και αρχίσουμε να γράφουμε συγκεκριμένα πράγματα για να βεβαιωθούμε ποιες είναι οι ανησυχίες των μεν και των δε. Για να προχωρήσουμε σίγουροι προς τη νέα νομοθεσία. Ξέρετε τη συνθήκη 10 φορές καλύτερα από μένα. διότι ήσασταν εδώ όταν τέθηκε σε ίσχυ και ξέρετε τι περιθώριο υπάρχει για την τακτική νομοθετική διαδικασία. Τη συνήθινη νομοθετική διαδικασία όταν μιλάμε για αυτόν τον τομέα. Ίσως όμως θα ήταν επικοδομητικό στο διάλογος να συζητήσουμε περαιτέρω για να γνωριστούμε καλύτερα για την υπόθεση Google. Νομίζω για μένα είναι, σαφέ, είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς την υπόθεση, να γνωρίζει τις απόψεις των άμεσα ενδιαφερομένων και για τα ένδικα μέσα της Google. Έχουν όλη τη γνώμη τους. Οι γνώμες έχουν εκφραστεί ήδη. Και είναι πολύ πτυχές οι απόψεις που έχουν εκφραστεί, το ίδιο και οι απαντήσεις και οι ιδέες γέννηκα μέσα της Google, οπότε πρέπει να περιμένουμε λίγο για να αποφασίσουμε για τα επόμενα βήματα. Αλλά όσο ευρύτερο το πεδίο, τόσο περισσότερα θέματα γύρονται και περισσότερο χρόνο θα χρειαστεί για να βρεθεί η λύση. Οπότε εδώ πρέπει να βρούμε μια, κάποια ισορροπία. Εάν θέλουμε όλα να λυθούν δια μιας, τότε θα χρειαστούμε πάρα πάρα πολύ χρόνο. Ο κύριος Κόφωτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και καλώ ήρθατε και πάλι, Επίτροπε, μετά την πολύ επιτυχημένη ακρόαση που είχαμε εδώ. Εκεί τονίσατε πόσο θεμελιώδους σημασία είναι για την Ευρώπη να έχουμε ελεύθερο και δίκαιο ανταγωνισμό. Μια δίκαιη πολιτική ανταγωνισμού. Θα επανέλθω στην υπόθεση των leaks ε, με τις διάφορες διαρροές. Εδώ είδαμε, αυτό να αφορά και άλλες χώρες, όχι μόνο το Λουξεμβούργο, ουσιαστικά κλέβουν εισόδημα από μια χώρα και το πάνε αλλού. Εάν δείτε τι έγινε το 2012, το κέρδος των Αμερικανικών πολυεθνικών ήταν 95 δις δολάρια όταν πέρναγαν μέσω Λουξεμβούργου. Και μόνο ένα δις κατέβαλαν σε φόρους. 1% φόρο από όλα αυτά τα χρήματα των Αμερικανικών πολυεθνικών που έχουν ε, δραστηριοποιούνται εδώ ε, στην άλλη πλευρά του Ελληνικού. Αυτό όμως συμβαίνει και μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών με τέτοιου φορολογικού παραδείσους. Αλλά και κάτι άλλο που είναι σημαντικό για να επανέλθουμε στη βάση του όλου θέματος είναι να υπάρχει δίκαιο ανταγωνισμός. Δηλαδή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να πληρώσουν 1% φόρο από τα εισοδήματά τους, τι να κάνουν. Αυτές δημιουργούν τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Αυτές χρειάζονται απεγνωσμένα στήριξη. Οπότε δεν μπορώ παρά να τονίσω κάποια από αυτά που ήδη αναφέρθηκαν. Οι ισχύοντες κανόνες ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι πολιτική ερώτησή μου, είναι επαρκή κατά τη γνώμη σα. Δείτε, τα, δείτε την πλευρά της δικαιοσύνης σε μια ε, ενιαία αγορά με κανόνες ανταγωνισμού, με ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, ανθρώπων και κεφαλαίων. Οι ίδιες χώρες κλέβουν εισόδημα η μία από την άλλη. Οι ίδιες χώρες που συμμετέχουν σε όλο αυτό. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Είναι σωστοί οι κανόνες. Είναι δίκαιες οι πολιτικές ανταγωνισμού. Και αυτές οι έμεσες κρατικές επιδοτήσεις που βλέπουμε με τέτοιου είδου φορολογικέ διευθετήσει. Δεν θα μπορούσαμε τουλάχιστον να συμφωνήσουμε εμεί ε, εμεί το Κοινοβούλιο και εσεί η Επιτροπή να πιέσουμε τα κράτη-μέλη. Ξέρετε πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα για κάποια κρατημέλη. Και το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία, ίσω κι άλλοι. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια πολιτική συμφωνία, να σταματήσει αυτού του είδου η πρακτική. Να υπάρχει δίκαιο ανταγωνισμό παντού. Ίσοι κανόνε παιχνιδιού για όλου. Ευχαριστούμε, Επίτροπος. Ναι. Αυτά που είπατε πλησιάζουν αυτά που είπε η, η Alice Και σας παρακολουθώ. Δεν έχουμε δύο διαφορετικές συζητήσεις που πολύ γρήγορα μπορούμε να τις περτέψουμε. Η μία είναι σαφής. Όταν έχουμε αποφάσεις για φορολογικά θέματα και υπάρχουν τέτοια. Είναι δίκες ή σε συγκεκριμένες αποφάσεις εμπλέκονται και θέματα ανταγωνισμού. Έχουμε κάποιες εκείνες υποθέσεις έχουμε γνώση, έχουμε νομική βάση. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούμε να αναλάβουμε δράση. Και όταν μπορούμε να αναλάβουμε δράση, θα πρέπει να το κάνουμε. Φυσικά θα πρέπει να ακούσουμε τα επιχειρήματα και των επιχειρήσεων και των ε, ενδιαφερομένων χωρών και μετά να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και επίσης έχουμε και θέματα φορολογικού ανταγωνισμού και φαινόμενα που είναι γνωστά και πάνω κάτω τα έχουμε αποδεχτεί. Υπάρχει δυνατότητα μεταθέσης χωρών από, με επιχειρήσεων από χώρες σε υψηλή προς με χαμηλή φορολογία. Πάντως είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσουμε την, τις προεργασίες που έχουν γίνει και την όθηση που έχει δοθεί στη συζήτηση για να περάσουμε στη συζήτηση του δεύτερου θέματος που είναι πιο λεπτό. Γιατί προϋποθέτει αλλαγές, πολιτική βούληση, πολιτικές αποφάσεις και ομοφωνία στο Συμβούλιο. Δεν είναι θέμα σύγκρουσης Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ή Επιτροπής και ε, Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να γίνει κοινή συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Γκούνερ Χοκμάρκ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καλώς ορίσατε, αγαπητή Δανέζα γειτόνισσα. Τι ερωτήσεις έχω να σας κάνω. Η πρώτη είναι, όταν συζητάμε για τις τράπεζες, είδαμε και θα δούμε και στο μέλλον ότι κάποιες τράπεζες θα πρέπει να κάνουν ανακεφαλαιοποίηση. Η κρατική ενίσχυση βοηθά. Όταν μάλλον υπάρχει κρατική βοήθεια χωρίς να υπάρχει επιστροφή χρηματών στο κράτος, είναι κρατική ενίσχυση. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς θα διασφαλίσετε ότι αυτό θα γίνει όταν θα γίνει ανακεφαλαιοποίηση των τραπέζων από τα κράτη στο μέλλον. Κάτι άλλο. Μου κάνει εντύπωση ότι μιλάμε για κρατική ενίσχυση. Όταν βλέπουμε τι προβάλλεται και στον τύπο, όταν προβάλλεται το θέμα του Λουξεμβούργου και ξεχνάμε την ευρύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά την κρατική ενίσχυση, τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, την ε, υπονόμευση της ενιαίας αγοράς. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξή. Προτίθεστε να δημιουργήσετε καταρχάς υψηλού επίπεδου διαφάνεια για το ποιος λαμβάνει κρατική ενίσχυση, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Είσαστε δεδεθειμένοι να προχωρήσετε με το στόχο της μείωσης του ποσού της κρατικής ενίσχυσης, γιατί μιλάμε πάντα για λεφτά φορολογουμένων που πληρώνουν διάφορες δραστηριότητες που πολύ συχνά στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Και υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, που μπορείτε να κάνετε αν επιδείξετε τόλμη στην θέση σας. Και νομίζω ότι έχετε τόλμη. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος ή Επιτροπός. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι και στο μέλλον θα υπάρξουν ε, ενδεχόμενες τράπεζες και, και περιπτώσεις τραπεζών που θα εξετάσουμε ενδεχόμενη ε, κρατική ενίσχυση. Γιατί παρά το γεγονός ότι θα υπάρξει η Τραπεζική Ένωση, η, η οδηγία για την εξυγίανση των τραπεζών, πάντα θα θέματα κρατικής ενίσχυσης. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε στην περίπτωση αυτή αν ακολουθούνται οι κανόνες, όπως είπα και προηγουμένως, σε ό,τι αφορά τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Εδώ λοιπόν θα διασφαλίσουμε ότι οι αρμοδιότητές μας στην Digicom θα μας επιτρέψουν να το ελέγξουμε αυτό και στο μέλλον. Είναι σημαντικό λοιπόν, πιστεύω, να συνεργαστούμε πολύ στενά με την ε, ενιαία εποπτική αρχή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να το πετύχουμε αυτό και ασφαλώς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Κατά δεύτερον, για την κρατική ενίσχυση και τη διαφάνεια. Νομίζω ότι ένα σημαντικό βήμα έγινε με τον εξυγχρονισμό της κρατικής ενίσχυσης, που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να δημοσιεύσουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν για την κρατική ενίσχυση. Όταν το κάνουν αυτό, υπό τον κανονισμό γενικών εξαιρέσεων. Αυτό δεν ήταν ε, αντιαφιλονίκητο, με το όλο έκανα εγώ, το έκανε ο προκατοχός μου, αλλά δεν ήταν κάτι το δεδομένο το αντιαφιλονίκητο Γιατί όπως είπατε, δεν, ήταν, ε, δεν είναι πάντα δεν είναι πάντα κάτι το δημόσιο, το τι έχει γίνει με τις δημόσιες δαπάνες, τα λεφτά των φορολογουμένων. Θα παρακολουθήσω την υπόθεση αυτή προκειμένου να πετύχουμε τη διαφάνεια αυτή που αποτελεί τον πυρήνα της ε, μεταρρύθμισης και να δούμε κατά πόσο υπάρχουν περαιτέρω βήματα που πρέπει να πάρουμε προκειμένου να επιτρέψουμε στους φορολογούμενους, στους πολίτες, στους εκλογείς να ελέγχουν το σκοπό για τον οποίο έχουν τα τα χρήματά τους. Ευχαριστώ λοιπόν ε, κύριε Επίτροπε, που ήρθατε να μας απαντήσετε στις ερωτήσεις σας και να ευχαριστήσω και τον κύριο Χουίκμαρ, ο οποίος μας επανέφερε στο θέμα μας επιτέλους. Αυτό θα το δείτε πολλές φορές εδώ, ότι φυσικά τα θέματα της καθημερινής πολιτικής επηρεάζουν και την ημερήσια διάταξη των συζητήσεών μας και τις τελευταίες ημέρες οι εφημερίδες δεν ανέφεραν τόσο πολύ τα stress test, αλλά μάλλον το θέμα της φορολογικής διαμόρφωση του συστήματο κάποιων κρατών μελών. Ένα άλλο θέμα να αναφέρω ότι χθε το Συμβούλιο οριστικά αποτέχτηκε την ε, πρότασή μα για τι δράσει αποζημιώσεων, μια πρώτη νομοθεσία με απόφαση όπου αποφασίζεται τι θα γίνει με το δίκαιο ανταγωνισμού. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα benchmark για τις μελλοντικέ δράσεις ε, Ελπίζω να ακολουθήσουν και περαιτέρω τέτοιε νομοθεσίε στην τρέχουσα θητεία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν κυρία Επίτροπε που ήρθατε και προσβλέπουμε στι μελλοντικέ ανταλλαγέ απόψε μαζί σα. Θα ήθελα επίση να περάσουμε στο 9, στα διάφορα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν, ε, ε αν υπάρχουν ε, παρατηρήσεις. Μάλιστα, επόμενη συνεδρίαση 17 Νοεμβρίου από τι 3 μέχρι τι 6.30 εδώ στι Βρυξέλλε. Σα ευχαριστώ και πέρα στη συνεδρίαση.